Gut, ich glaube, wir können dann starten und zwar... Αρχίζουμε, αρχίζουμε. Ορίζοντας 2020 ελαφρά οχήματα, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα από τις εκπομπές των ε, ελαφρών οχημάτων. Εντάξει, δεν φτάνει εδώ απλή πλειοψηφία. Ψήφισαν όλοι. Μάλιστα. Πέρασε. 37 υπέρ 5 κατά καμία αποχή. Εντάξει, ε, εγκρίθηκε αυτή η νομοθετική διαδικασία και προχωρούμε. Σημείο 10. Είναι για τα απόβλητα από χαρτί ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 34 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά. Δεκτό και αυτό. Πάμε παρακάτω. Σημείο 11. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά Απόβλητα. Το έχουμε αναβάλει μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων αυτή ε, θα ψηφιστεί τέλος Νοεμβρίου, είναι του Βιτόριο Πρόντι. Στις 27 ενδεκάτου συγκεκριμένα, τότε θα ψηφίσουμε αυτή, αυτό το θέμα. Ε, συνάδελφε Μπονανίνη, σημείο 12, αρχίζουμε πρώτη ψηφοφορία, 55 τροπολογία σε τρία μέρη. Πρώτο υπέρα Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ε, δεκτό. Τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό και αυτό. Καταπίπτει 57 και συνεχίζουμε με την 56 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58 και 59 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεκτές 7 και 60 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές ψήφισαν μόνο φιλελεύθεροι και πράσινοι δεν φτάσαμε στην απαρτία στην πλειοψηφία που θέλαμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία Εψήφισαν όλοι πέρας σαφώς δεκτές. Οι μεγάλες ομάδες παρακαλούνται να μην αφήνουν να δουλεύουν μόνο οι μικρές. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 62 και 64 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 65 και 66 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Είχε απορριφθεί εκείνη. Η συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καταπίπτει 15. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφέ Ελέγχουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 74 άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 75-76 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτέ. 77 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 19 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 80. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Με ισχνή πλειοψηφία. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές ασαφές. Ψηφίζουμε την 21 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή, 94 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, 30. Α, έλεγχος, έλεγχος, στην 95. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. 30 και 96 ταυτόσημες. Πέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές απορριπτέται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Ε, συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 104 υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε την 104 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός 337. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 39 σε δύο μέρη. Ένα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 και 109 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τη 41. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Όχι, δεν πρέπει να, το ψηφί, την ψηφίσουμε αυτή, γιατί δεν έγινε δεκτή η 95. Να ψηφίσουμε, λέτε. Α, ε, να ψηφίσουμε. 42, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. Πάμε στη 43 υπέρ. Κατά. Αποχές Ασαφέ Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 43 άκρη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 112 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 113 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός 113. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία, 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 47 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 48. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Σαφώς δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 και 51 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά ασαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 53 άρχεται ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή καταπίπτει οι δύο ψηφίζουμε την 3 και την 54 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 51 ψήφι υπέρ, 0 ψήφι κατά, 0 αποχές. Ε, θερμά συγχαρητήρια κύριε Μπονανίνη. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ψηφοφορίες και Τώρα περνάμε στην έκθεση της συναδέλφου Λίντα. Α, α, α, είχαμε πει για μία αλλαγή στη σειρά. Ναι, πρώτα είπαμε ότι θα ε, πιάσω με την έκθεση του κυρίου Ρώση και μετά της κυρίας Μακάιβαν. Οπότε δίνω πρώτα Αφού επικρατήσει ησυχία, δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρώση. Ορίστε κύριε Ρώση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση αρκετά πολύπλοκη γιατί είναι τεχνική και αφορά την προστασία απέναντι σε επιβλαβείς οργανισμούς για τα φυτά που βρίσκονται μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σπόρους και φυτά που εισάγονται από το εξωτερικό. Και μιλάμε για συστήματα και μεθοδολογίες για την εκρίζωση των ε, ε, ε, οργανισμών αυτών ή για το πώς μπορούν να θεραπευτούν τα φυτά που έχουν προσβληθεί. Τα μέτρα αυτά χρησιμεύουν για την βιωσιμότητα της γεωργίας και για την ε, βελτίωση ε, της εισαγωγής ε, νέων φυτών, ίσως ανθεκτικών, για την οικηβευτική και την δασοκομεία και την γεωργία και για την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων μας. η γεωργία, η κυπευτική και η δασοκομεία μας απειλούνται από νέα παράσιτα με μεγάλες επιπτώσεις και για την υγεία των φυτών αλλά και των προϊόντων των φυτών και όλο αυτό σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και τις κλιματικές αλλαγές. Ε, δέχομαι ευνοϊκά την πρόταση αυτού του κανονισμού για την ε, ε, προστασία που έχει σαν σκοπό ε, την ε, καλύτερη αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν και αμφιβολίε όσον αφορά τι μεθόδου που θα χρησιμοποιηθούν, έστω και αν είναι θεμητέ. Παραδείγματο χάρη, σχετικά με τις προτεραιότητες που δίνονται. Δεν είναι λανθασμένο ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι τα φυτά που πιθανόν να έχουν προσβληθεί θα πρέπει πρώτα να ελέγχονται και μετά να εκριζώνονται. Γιατί αυτό αν δεν γίνει παραμένουν οι αιστείες και υπάρχει κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας ε, και μην ξεχνάτε το περίφημο ε, σκαθάρι ας πούμε που αν το ε, αφήσω θα ε, διαδοθεί αλλού. Τώρα για την πρόταση, σε γενικές γραμμές συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να περάσουμε σε λεπτομέρειες για ορισμένε συγκεκριμένε πτυχέ, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κατάλογο των επιλογών οργανισμών και την, και την ε, ανάγκη ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση και όχι εκτελεστικών πράξεων. Στην πρόταση η Κομισιόν προτείνει πάρα πολλέ εκτελεστικέ ε, πράξει ε, που αφορούν τον κατάλογο επιλογών οργανισμών καραντίνας. Τα, οι επιλογές οργανισμοί προτεραιότητας, δηλαδή οι οργανισμοί για τους οποίους θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, αυτοί δηλαδή που είναι οι πιο επικίνδυνοι, η πιο χώρο κατα... Ε, μιλάμε επίσης για τις προστατευόμενες ζώνες, προστατευόμενες ζώνες καραντίνας και ε, τους οργανισμούς που βλάπτουν την ποιότητα. Για όλες αυτές τις διατάξεις πιστεύω ότι οι πράξεις εξοδότηση είναι το καλύτερο μέσο ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι δίνεται έτσι στο κοινοβούλιο, δίνονται στο κοινοβούλιο οι απαραίτητες εξουσίες για να ε, τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους καταλόγους αυτούς. Θέλω να ακούσω και εσάς και ιδιαίτερα τους σιώδεις συζητητές όμως αν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να δώσουμε το ελεύθερο στην Κομισιόν. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο να διατηρήσει τις εξουσίες του και το Κοινοβούλιο. Ε, προτείνω λοιπόν τροποποίηση του άρθρου 98.2 που αφορά ακριβώς αυτό το θέμα της πράξης κατεξουδότηση ε, και αυτό με διάρκεια 5 ετών, η στάντα ρήτρα δηλαδή. Μετά, το άλλο επίμαχο σημείο είναι ο περιορισμένος αριθμός ε, επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας. Δηλαδή αυτή που είναι πιο επικίνδυνη. Η Κομισιόν προτείνει αυτό να είναι το 10% του αριθμού των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας. Οι επιβλαβείς οργανισμοί ε, προτεραιότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί έχουν, ε, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό για την επικράτειά μας. Ε, χρειάζονται μεγαλύτερη ε, ετοιμότητα αντίδρασης, ετοιμότητα των φυτογενικών υπηρεσιών αλλά και των τοπικών αρχών όταν πρέπει να επεμβαίνουν και μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι ο ρυθμό των ε, παρασύτων δεν πρέπει να είναι περιορισμένο, αν θεωρούνται πραγματικά ε, επικίνδυνα. Αν υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις ε, επικίνδυνων επιλαβών οργανισμών, γιατί θα πρέπει ο ρυθμός να περιοριστεί στο 10% του συνόλου. Αν είναι περισσότερα αυτά τα παράστα μπορεί να είναι 20-30%. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό ο περιορισμό. Ενημέρωση του κοινού. Το θέμα εδώ είναι η πλήρης, σχεδόν πλήρη έλλειψη τη ενημέρωση του της κοινή γνώμη, για τον κίνδυνο που ε, ε, έχουν οι επιβλαβείς αυτοί οι οργανισμοί. Ε, όχι μόνο για την υγεία των φυτών, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό προτείνουμε Προτείνονται καμπάνιε ευαισθητοποίηση στο επίπεδο των κρατών μελών ώστε να ενημερώνονται οι πολίτε για του κινδύνου που σχετίζονται με την εισαγωγή φυτών από τρίτε χώρε. Και επίση και για τα φυτά που αγοράζονται μέσω του διαδικτύου η Κομισιόν θα πρέπει να διαθέτει στο κοινό ένα επικαιρωμένο κατάλογο ε, των παρασίτων από τρίτες χώρες και από αναδυόμενες χώρες για τους κινδύνους που ενέχουν για την ε, υγεία των φυτών αλλά και για την ε, δημόσια υγεία. Ε, διαδικτυακό εμπόριο, άλλο πρόβλημα. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αυτό το εμπόριο μπορεί να αποτελεί ένα ψηλό κίνδυνο φυτογενομικό, διότι τα εμπορέματα αυτά μπορεί να είναι από ε, αλόχθονες επιβλαβείς οργανισμούς, ε, ε Πρόκειται λίγα δηλαδή παράσιτα που σήμερα ε, για τα οποία μάλλον σήμερα δεν υπάρχουν ε, επαρκή τρόποι αντιμετώπιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χρειάζεται η καραντίνα. Ιδιαίτερα η εισαγωγή φυτών από τρίτε χώρε που αγοράζονται μέσω του διαδικτύου πολλέ φορέ δεν ε, συμμορφώνονται με του φυτογενικού κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των εμπόρων λοιπόν φυτών θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον ευαισθητοποίηση προτείνουμε να να ενισχυθεί η πρόταση της Κομισιόν προσδιορίζοντας ότι οι διαδικτυακοί έμποροι δεν μπορούν κατά κανέναν τρόπο να εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφή σε Μητρό. Τελειώνω σχεδόν, Πρόεδρε. Συμμετοχή των δεδομένων μερών στην εκπόνηση σχεδίων έκθεση ανάγκη και ασκήσεων προσωμείωση. Η συμμετοχή όλων αυτών ποικίλει σήμερα από κράτος σε κράτος. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για την έγκαιρη συμμετοχή των επαγγελματιών σε αυτά τα είδη δραστηριοτήτων. Τελευταίο σημείο, χρηματοοικονομικές πτυχές, θα πρότεινα δύο σημαντικές τροποποιήσεις στο άρθρο 102. Πρώτον, η πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση δαπανών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την πρόταση για την πρόληψη και την διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών και να επιτρέπει τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα όσον αφορά τις δαπάνες που υφίσταται τα κράτη-μέλη για την αποζημίωση ε, των ε, καλλιεργητών που θα είναι ίση προς το κόστος των καταστραφέντων φυτών. Και ένα άλλο θέμα που πάλι σχετίζεται με το οικονομικό, ε, Αυτές οι έγκαιρες πράξεις είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την ανείχνευση και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας και γι' αυτό τα αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας που εκτελούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις, για αποζημιώσεις. Δηλαδή όταν υπάρχουν ε, οι ιδιώτες ή ε, δημόσιοι φορείς που είναι υποχρεωμένοι να εξεριζώσουν κάποιες ε, ε, καλλιέργειες, κάποια φυτά, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται αποζημίωση για να αποζημιώνονται ε, επιχειρήσεις που χαρίζει καμία δικιά τους ευθύνη βρίσκονται με χωροκρατικά παράσιτα και επιλογή οργανισμούς μέσα στις καλλιέργειες τους. Αυτά πρόεδρε και όπως σας προειδοποίησα είναι αρκετά τεχνικός ο κανονισμός. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Ρώση. Ε, κυρία... Κύριος... Κυρία Σάμπορφ έχει το λόγο. Ε, Σκιώδης. Κυρία Σάρμπου. Εγώ θα διαβάσω αυτά που έγραψε ο συνάδελφος, κυρίως Δαναμπρέσκου, που δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, Πρέπει να δράσουμε γρήγορα στα πλαίσια της στρατηγικής ε, για τα, τους επιβλαβείς οργανισμούς γιατί και η γεωργία και άλλοι τομείς ε, βλάπτονται. Ε, συγχαίρω τον συνάδελφο Ρώση για τη δουλειά του. Συμφωνώ με τις περισσότερες ε, προτάσεις σε σχέση με την έγκριση κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, για τη θέσπιση καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών. Χρειάζεται και μία ενημέρωση της κοινή γνώμης για ενδεχόμενους κινδύνους από επιβλαβείς οργανισμούς. Όμως δεν συμφωνώ ότι μόνο οι ειδικοί θα πρέπει να ενημερώνονται όταν πρόκειται για προσωμείωση και έκτακτη ανάγκη. Στο 22 και 24 σημεία. Εκεί νομίζω ότι είναι πολύ περιοριστικό το κείμενο γιατί πρέπει να λαμβάνονται και άλλοι παράγοντες υπόψη με τις διαδικασίες εκτάθης ανάγκης και στο 19 εκεί τα κράτη-μέλη και οι γεωργοί έχουν την δυνατότητα, τις τροπολογίες αναφέρομαι, ε, ε, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ε, τα απαραίτητα μέτρα. Νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε και μέσα από το περιβαλλοντικό πρίσμα και όχι μόνο μέσα από το οικονομικό πρίσμα και την κερδοφορία. Ε, έτσι θα προστατεύεται καλύτερα το περιβάλλον. Ε, επίσης από την πρόταση της Κομισιόν λείπουν ε, και μέτρα κατά κινδύνων απελευθέρωσης τέτοιων επιβλαβών οργανισμών ουσιών. Και πρέπει ακόμη να φροντίσουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ε, λειτουργούν με βάση την αρχή της προφύλαξης και να προστατεύεται και η δημόσια υγεία και το περιβάλλον παράλληλα. Θα πρέπει να προβλέψουμε δημοσιονομικά εξισωτικά ποσά για, ως αντισταθμίσεις από όλους όσους ε, εργάζονται σε αυτό το τομέα θα πρέπει να επιληθούν θέματα ε, το άρθρο 73 και 77 είναι σχετικά για την έγκριση συγκεκριμένων επαγγελματιών μέσα από την έκδοση των διαβατηρίων. Είναι το άρθρο επίσης 84 που θα πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Ακόμα λείπει ένα συνολικό, μια συνολική θεώρηση ε, αυτών των επιβλαβών οργανισμών στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στην κειμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τώρα ο Τζέιμς Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ. να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά που έκανε στα πλαίσια της γνωμοδότησης και περιμένω να συνεργαστώ τις επόμενες εβδομάδες μαζί του πάνω σε αυτό το φάκελο για να βρεθούν καλές συμβαστικέ λύσεις. Είναι σημαντικό να γίνονται πιο αυστηροί έλεγχοι σε, αυτή την, σε αυτό το τομέα γιατί το προηγούμενο χρόνο είδαμε ότι οι χαλαροί έλεγχοι οδήγησαν σε καταστροφικά αποτελέσματα γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε έξαρση νόσου που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα στη χώρα μας μέσα από τα ε, νοσούντα φυτά. Χρειάζεται ευελιξία για αποτελεσματικότητα, χρειάζεται προερόληψη και γρήγορη δράση για την προ... Ε, παρεμπόδιση της εξάπλωσης της νόσου. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν μέσα από τη, το καινούριο, την καινούρια πρόταση. Ε, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες εις ό,τι αφορά τα παράσιτα. Θετικό είναι αυτό καταρχήν, γιατί μας βοηθάει να επικεντρώνουμε στους πόρους και τις δράσεις. Είναι σαφές ότι η στοχοθέτηση θα δουλέψει στην πράξη και θα λάβει υπόψη και κλιματικά και γεωγραφικά κριτήρια και διαφορές και εθνικές ανάγκες και θα αντιμετωπίσει νέους πάλι και νέους και πάλι επανερχόμενους κινδύνους. Θα πρέπει να ορίσουμε τους κινδύνους και τα παράσιτα. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις στο παράρτημα της πρότασης. Ε, ε, είναι καλύτερο να είμαστε συγκεκριμένοι και να μην έχουμε αυθαίρετο περιορισμό 10%. Επίσης καλό είναι να ε, αναφερθούμε στις ε, εκτελεστικές και τις κατεξουσιοδότηση ε, σε ό,τι αφορά στην, ε, τον κατάλογο των παρασίτων. Αυτό είναι πρόβλημα που αφορά όλο το πακέτο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το ζήτημα των πράξεων σωστά και να κάνουμε και τις απαραίτητες προσαρμογές στις διαπραγματεύσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αυθυγραμμίσουμε την πρόταση κανονισμού σε διαχείριση των δαπανών σε σχέση με την πρόταση της ε, Κομισιόν για τα ξένα είδη. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει τη δουλειά της πάνω σε αυτό το φάκελο και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν από την επόμενη Ολομέλεια και πριν από τις εκλογές. Ε, μπορεί να ε, ανοίξουν τα θέματα στα πλαίσια των συζητήσεων με το Συμβούλιο. Εμείς θα πρέπει να έχουμε έτοιμη την νομοθεσία μέχρι τον επόμενο Απρίλιο. Δεν συμφωνώ με την πρόταση αναθεώρησης των δομών όπου λέει ο εισηγητής ε, για να δοθεί ε, πληροφορία στο κοινό. Ε, θα πρέπει να γίνει πιο ε, συγκροτημένα και να μην ε, παραμελούμε το, τα κράτη-μέλη και να επικεντρώνουμε μόνο στις ε, τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω με χαρά να συνεργαστώ με τον ε, εισηγητή. Τέλειωσαν οι εισηγητές. Η Κρίστα Κλάς τώρα και μετά η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ορέστερό για την έκθεση και Τώρα πια επιτέλους μιλάμε και για την υγεία των φυτών, γιατί πριν από λίγα χρόνια την οδηγία για την προστασία των ε, φυτών την είχαμε περιορίσει στα παράσιτα. Τώρα μιλάμε και γενικότερα για την υγεία που προϋποθέτει διατήρηση, διαφύλαξή της και από την άλλη όταν υπάρχει νόσος θα πρέπει να καταπολεμείται. Ε, πρέπει να προσέξουμε βέβαια να υπάρχει ε, συνοχή μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών. Ε, πρόληψη, καταπολέμηση και έχουμε και νέους επιβλαβείς οργανισμούς γιατί είχαμε θερμ... υψηλές θερμοκρασίες τα προηγούμενα χρόνια. και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, γιατί έχουμε την αρχή της προφύλαξης ε, που είναι πολύ σημαντική. Ε, είπαμε ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε και την έρευνα και θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ρωτήσω και την Κομισιόν σε ποιο βαθμό προχώρησε η υλοποίηση ε, εντατικοποίηση της έρευνας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών ουσιών για καλλιέργειες, που θα στηρίζονται στην αρχή του minor use, ε, μικρότερη χρήση. Ε, εκεί δεν έχει προχωρήσει ακόμη η Κομισιόν. Ε, Επίση ε, μιλούσαμε και για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Τώρα επανέρχεται στο θέμα αυτό ο συνάδελφος Ρώση. Λοιπόν πρέπει να δούμε ε, και να ρωτήσουμε εδώ τι γίνεται με την υλοποίηση γιατί είχαμε πει ότι θα γίνει το 2014. Έφτασε το 2014. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της φυτοπροστασίας. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό. Επίσης συνάδελφε Ρώση, το κατάλογο των προσδήλωση επιβλαβών οργανισμών πρέπει να περιοριστεί στο απαραίτητο. Κάθε επιβλαβής δηλαδή οργανισμός που δηλώνεται συνεπάγεται πληθώρα γραφειοκρατίας και ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί που δεν επεκτείνονται, δεν πολλαπλασιάζονται πολύ, ίσως δεν πρέπει να ε, δηλώνονται. Ε, να ρωτήσουμε και τους επιστήμονες, αλλά καλό θα ήταν να, να περιοριστούμε στους σημαντικούς οργανισμούς. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούζο. Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Και συμφωνώ με αυτά που άκουσα. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό τώρα μέσα σε μια νομοθετική πράξη να συμπεριλάβουμε όλα αυτά που αναφέρθηκαν και που αποτελούν μέρος ενός γενικότερου φυτογενομικού πακέτου. Κάτι το οποίο απλοποιεί, εναρμονίζει, διευκολύνει τον χειρισμό των θεμάτων αυτών. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε για την πρόταση αυτή είναι ότι πρόκειται για κάτι αρκετά γενικό και λείπουν συγκεκριμένα ζητήματα. Ο κανονισμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία, τα σημαντικά, χωρίς να δίνει τόσες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση πράξη είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό, αλλά παραμένουν πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα ακόμα ανοιχτά. Όπως επίσης ο κατάλογος για την καρατίνα, τα προστατευμένα φυτά και οι αντιστοιχίες. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην βασική νομοθετική πράξη. Όπως επίσης οι επιδημίε είναι επίση κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρεται εδώ. Υπάρχουν διαφορετικές βέβαια απόψεις όσον αφορά τον κίνδυνο, ε, διαφορέ απόψεων ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ μιας πιο πλήρης προσέγγισης. Αυτός ο κατάλογος κατά προτεραιότητα ε, πρέπει να ορίζεται πολύ καλά στον νέο κανονισμό. Προτείνουμε επίσης το ανώτατο όριο να διαγραφεί. Γιατί πιστεύουμε ότι ο αριθμός αυτός προτεραιοτήτων εξαρτάται από τον κίνδυνο και εξαρτάται από τη σημασία που έχει ανάλογα με την περιοχή της Ευρώπης την οποία εξετάζουμε. Χρειάζεται επίσης και διευκρίνηση για την δυνατότητα δράσεων σε ιδιωτικές μονάδες εγκαταστάσεις. Το λέω αυτό γιατί ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβουμε εγκαταστάσεις, κατοικίες ε, ιδιωτών. Όσον αφορά τώρα τις προστατευμένες περιοχές, το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή δεν επιτρέπει μετακίνηση ε, φυτών από μία ε, περιορισμένη περιοχή. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να μην είμαστε τόσο απόλυτοι, ας το εξετάσουμε περισσότερο αυτό. Στην περίπτωση του υλικού δηλαδή που προέρχεται από περιοχές μη προστατευμένες. Ο κανονισμός επίσης αφήνει εκτός πεδίου τα Κανάρια και κάποια γαλλικά επερπόντια διαμερίσματα. Αυτό πρέπει να το μελετήσουμε γιατί υπάρχουν επιπτώσεις και γίνεται σημαντικό εμπόριο φυτών από τις Κανάριες νήσους προς την Ευρώπη. Γι' αυτό τα Κανάρια δεν θα πρέπει να μείνουν εκτός κανονισμού. Όσον αφορά τώρα τους επίσημους ελέγχους, εδώ χρειάζεται αύξηση του προσωπικού, του καταρτισμένου προσωπικού με προσόντα. χρειάζονται, όπως είπαμε, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε λοιπόν ο κανονισμός να καθορίζει τις γενικές προϋποθέσεις, τις βασικές προϋποθέσεις και τα κράτη-μέλη να είναι εκείνα τα οποία θα αποφασίζουν για το ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Δεν είμαστε κατά της αγόρευσης να υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση δεν υπάρχει σχέση με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό που συζητάμε αυτή την εποχή, μέσω του οποίου καθορίζονται δημοσιονομικές προδιαγραφές για τους φυτογενομικούς κανόνες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να ξέρουμε τη σχέση μεταξύ των δύο κανονισμών για να μπορούμε και να αξιολογήσουμε τελικά ποιες περιπτώσεις θα επιδέχονται χρηματοδότηση και ποιες όχι. Κάρεν, ευχαριστώ. Δυο σκέψεις ε, θέλω να κάνω. Ε, αρχή προφυ... που αναφέρονται στην αρχή προφύλαξης και τη σύνδεση με την ΚΑΠ. Δεν πρόκειται μόνο για καταπολέμηση μέσα από παρασιτοκτόνα, αλλά το θέμα είναι γενικότερο και αφορά τη διεξαγωγή της γεωργίας που θα πρέπει να περιλαμβάνει περιβαλλοντικά μέτρα, αμυψή σπορά ε, και άλλα που καταπολεμούν τους επιβλαβείς οργανισμούς. Νομίζω ένας τέτοιος κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την εναλλακτική γεωργία. Ε, μέσα από τις μονοκαλλιέργειες και ακριβώς την ίδια ε, καλλιέργεια προάγεται και ο πλαπλασιασμός των επιβλαβών οργανισμών. Ε, τότε θα καταπολεμήσω ή μήπως πρέπει να ε, στραφώ περισσότερο στην εναλλακτική γεωργία όπου χρειάζομαι και πολύ λιγότερα παρασιτοκτόνα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε αυτόν τον προβληματισμό. Ευχαριστώ την Κάρεν Κάντενμπαχ και τώρα η Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος? Όχι. Υπάρχει, υπάρχει. ο εκπρόσωπος, ο κύριος Πόλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά τους στο έργο αυτό, που λαμβάνουν υπόψη τους πολλές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αναφερθώ σε διάφορες πτυχές που ανέφεραν και μέλη της Επιτροπής σας. Το πρώτο έχει να κάνει με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ή τις εκτελεστικές. Κοιτάξτε, εδώ βρισκόμαστε βέβαια στον πυρήνα της διοργανικής συζήτησης ανάμεσα στο Συμβούλιο, τη Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και έχουμε παρακολουθήσει τι λέει η συνθήκη της Λισαβόνας που προτείνει ότι ο κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών τροποποιείται μέσω εκτελεστικής πράξης. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ βαρύ όμως να μπει κάτι στο σημερινό κείμενο, γιατί ο κατάλογος αυτός ε, τροποποιείται τακτικά μέσω γρήγορων διαδικασιών, κάθε φορά δηλαδή που εμφανίζεται μια νέα ασθένεια για παράδειγμα. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε εκτελεστική πράξη. Δεύτερον, οι αποζημιώσεις οικονομικές, τις σταθμίσεις. Είναι σημαντικό γιατί βλέπετε η δράση μας στρέφεται γύρω από τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι γρήγορη κοινοποίηση από τους παραγωγούς με άμεση διάγνωση για να καθορίσουμε ποια είναι η ασθένεια εδώ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι γρήγορα μέτρα από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο τρίτος πυλώνας είναι οι οικονομικές αποζημιώσεις ανάλογα με την ζημιά που έχει προκληθεί από τους επιβλαβείς αυτούς οργανισμούς ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν πολύ γρήγορα να κοινοποιούν. Δυστυχώς έχουμε παραδείγματα κοινοποίησεων που έγιναν στις εθνικές αρχές ένα χρόνο, δύο χρόνια και τρία χρόνια ακόμα αφού εμφανίστηκε το πρόβλημα επιτόπου. Όταν λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι ο επιβλαβής οργανισμός διαδίδεται, ε, μεταφέρεται και καλύπτει μια πολύ μεγάλη πια επιφάνεια, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν μέτρα εκρίζωσής του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, είτε πρόκειται για δασοκόμη, είτε αγρότε, ε, οτιδήποτε, να είναι πολύ γρήγοροι στην κοινοποίηση. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η οικονομική αυτή αποζημίωση. Και όχι μόνο για τα σχέδια δοκιμών, αλλά και για την εκρίζωση δέντρων, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υποχρεώνουμε ε, ο παροφόρα δέντρα να τα κόψει ο ιδιοκτήτης τους, όπως έχει γίνει με τις πορτοκαλιές στη Σικελία, καταλαβαίνετε ότι η ζημιά είναι μεγάλη. Ε, φυτεύεται ένα καινούριο δέντρο, το οποίο δίνει όμως πορτοκάλια μετά από 5-10 χρόνια. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, ο ιδιοκτήτης δεν έχει έσοδα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το πλαισιώσουμε φυσικά για να μην γίνονται καταχρήσεις. Δεύτερον, ενημέρωση του κοινού. Αναφέρθηκαν πολλοί εδώ στην Επιτροπή σας αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό το κοινό να ενημερώνεται, ιδιαίτερα για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Στα αεροδρόμια όλοι βλέπουμε τις αφήσει που υπάρχουν και που προειδοποιούν ότι απαγορεύεται εισαγωγή γάλακτος, κρέατος κτλ. οι αφήσει αυτές θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από διπλές αφήσει. Να υπάρχει μία για τα ζωικά προϊόντα και μία για τα φυτικά. Γιατί οι τουρίστες μπορούν να φέρουν ε, φρούτα ή μικρά γλαστράκια με φυτά, χωρίς να το ξέρουν, να προκαλέσουν ασθένειες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Είναι επίσης σημαντικό, το αναφέρατε κι εσείς, ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει στις ασκήσεις έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξέρουμε και να βλέπουμε πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν οι αρχές. Εννοείται. Τώρα θέλω να πω και δύο λόγια για τα χωροκατακτητικά είδη. Είναι και αυτό σημαντικό. Ξέρετε ότι οι συνάδελφοί μας από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος πρότειναν ένα κείμενο για τα χωροκατακτητικά αυτά είδη φυτά και ζώα. Τη χρηματοδότηση πρέπει να τη δούμε σε αυτό το πλαίσιο, όμως και όχι στα πλαίσια της υγείας των φυτών. Επόμενο σημείο. Πολλέ φορές αναφέρθηκε η πρόσβαση ε, στους ιδιώτες όταν δέντρα, φυτά πλήττονται από κάποια ασθένεια. Εννοείται, επίσημες υπηρεσίες δεν πρόκειται να μπαίνουν στους κήπους των ανθρώπων χωρίς να τους ενημερώνουν, δεν θα πηγαίνουν να κόβουν, να καταστρέφουν φυτά, δέντρα, μερικές φορές μεγάλης αξίας, όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά είναι σημαντικό, εφόσον έχει διαγνωστεί μια ασθένεια στον ιδιωτικό χώρο, σε ένα κήπο, σε ένα πάρκο, σε ένα γκολφ, σε ένα γήπεδο του γκολφ. Οι φυτογενομικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να παρέμβουν για να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα, είτε να θεραπεύσουν τα φυτά που έχουν πληγεί από την ασθένεια, είτε πολλές φορές χρειάζεται να τα κόψουν, να τα καταστρέψουν, προκειμένου να μην αποτελέσουν εστία ασθένειες που θα μεταδοθεί ε, και πιο πέρα. Αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να την έχουμε, αλλά εννοείται ότι πρέπει να πλαισιώνεται η δυνατότητα αυτή και πάλι για να αποφεύγονται καταχρήσεις. Θέλω να απαντήσω και στην κυρία Κλάς τώρα για τα παρασιτοκτόνα μια που δεν αποτελεί το θέμα αυτό αντικείμενο της έκθεσης αυτής ούτε του κανονισμού. Για τα φυτογενομικά αυτά προϊόντα, τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο, για τα ζώα, τα έντομα, για το περιβάλλον, πολλές φορές απαγορεύονται. Θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται για μικρά είδη σε περίπτωση αιστιών. Υπάρχει δυνατότητα στην φυτογενομική ρύθμιση σε περίπτωση εστιών νέων ασθενειών που εμφανίζονται να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρασιτοκτόνα τα οποία οι υποκανονικές συνθήκες δεν επιτρέπονται. Και αυτό για να θεραπεύσουμε φυτά για τα οποία δεν προορίζονται κανονικά τα παρασυτοκτόνα αυτά. Η κυρία Κλάς Αναφέρθηκε επίσης στην οδηγία για την ε, ολοκληρωμένη προστασία των φυτών που θα αρχίσει να ισχύει το 2014. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία και έχουμε συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εγκαθιδρύσουν τα αναγκαία μέτρα, ιδιαίτερα την κατάρτιση των αγροτών, να τους ευαισθητοποιήσουν ε, στους κινδύνους που υπάρχουν από τη χρήση φυτογενομικών προϊόντων, ε, τιμένοι πάνω στο φυτό για τους κινδύνους στο περιβάλλον που περνάνε πολλές φορές στα υπόγεια ύδατα ή στα ποτάμια. Έπειτα να δούμε και τη ρύθμιση των ε, μηχανών που ψεκάζουν ε, τα προϊόντα αυτά. Να περιοριστεί η ποσότητα του ύδατος για παράδειγμα. Δουλεύουμε πάνω σε όλα αυτά μαζί με τα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε μαζί τους και σε πολλές χώρες έχει προχωρήσει το θέμα πολύ. Θέλουμε και μια έκθεση ενημερωτική για την εφαρμογή και θα την έχουμε στους επόμενους μήνες. Τώρα για την εκπεριτροπής ε, καλλιέργεια φυτικών ειδών. Τώρα όλοι οι πυρογνώμονες, είτε είναι γεωπόνοι, είτε είναι φυτογειονομικοί, συμφωνούν και λένε ότι αυτή η εκπεριτροπής καλλιέργεια είναι μια πρακτική αναγκαία για να βελτιωθεί η απόδοση των γιών και για να μειωθούν οι επιπτώσεις των ασθενειών. Είναι προφανές ότι όταν για πάρα πολλά χρόνια στον ίδιο χώρο, στο ίδιο αγροτεμάχιο έχουμε την ίδια καλλιέργεια, εξαντλείται γεωπονικά το κομμάτι αυτό της γης, άρα χρειάζονται περισσότερα λοιπάσματα, άρα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες μετάδοσης ασθενειών μέσω βακτηριδίων κλπ. Όλοι οι συμφωνούν για την εκπεριτροπή σε αυτή καλλιέργεια, διαφορετικές καλλιέργειες δηλαδή στο ίδιο αγροτεμάχιο. Υπάρχει ένα έντομο, το σέκτικα για παράδειγμα, το οποίο θέλουμε να το καταστρέψουμε και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το να επιβάλλουμε αυτή την πρακτική, οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας δεν το θέλουν στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής, το υποχρεωτικό δηλαδή. Θέλουμε όμως και εμείς και εκείνοι να δίνουμε κίνητρα, να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να χρησιμοποιούν αυτήν την εκπεριτροπής διαφορετικές καλλιέργειες στα αγροτεμάχια τους. Αυτά είχα να απαντήσω στον εισηγητή και στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ρώση θα πάρει το λόγο για να συνοψίσει και να κλείσει το θέμα. Ορίστε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι άνοιξε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ και εγώ όλους τους συναδέλφους, τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές και την Κομισιόν. Συμφωνώ ότι για τα παρασιτοκτόνα είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει ανοχή ε, στους ζυζανικτών εκ μέρους των ε, επιβλαβών οργανισμών. Ιδίως για τα εσπεριδοειδή ε, είδαμε ότι τα παλιά ζυζανικτόνα είναι σχεδόν άχρηστα πλέον. Άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ε, ότι όντως ε, η συνάδελφος έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να προβλέπεται ένας ολοκληρωμένος πόλεμος κατά των επιβλαβών οργανισμών στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ε, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα της ε, πράξης κατεξοδότησης ή εκτελεστικής πράξης, ε, είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε ε, αρκετά γρήγορα ε, όταν μας θέσει τα σχετικά ζητήματα η Κομισιόν. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή καθυστέρησης λόγω της πράξης κατεξοδότηση. Ε, τώρα, για όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε ε, μια κοινή γραμμή αγώνα κατά των επιβλαβών οργανισμών και κατά την εισαγωγή τους και να υιοθετήσουμε τις βέλτιες πρακτικές και για την την πιθανή θεραπεία των προσβεβλημένων φυτών. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να ενεργούμε ταχύτατα και εκτιμώ επίσης αυτό αυτά που υπόθηκαν για τον κατάλογο των ε, οργανισμών ε, που θα πρέπει να κοινοποιούνται. Ε, ναι, ναι, είναι περιορισμένος αυτός ο κατάλογος, αλλά γιατί να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι περιττό. Ε, βεβαίως όσο περισσότεροι οργανισμοί περιλαμβάνονται τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. Για την ενημέρωση τώρα σχετικά με τα πιστοποιητικά για τα φυτά, ε, συμφωνώ για το θέμα του ίντερνετ, ε, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και όπως είπε και η Κομισιόν, η ενημέρωση πρέπει να δίνεται στα σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λιμάνια, ε, αεροδρόμια κλπ, ώστε να υπάρξει πρόληψη. Τώρα, συμφωνώ και ευχαριστώ την συνάδελφο Αγιούζο, που ε, είναι πρόθυμη να αρχίσει να εργάζεται για το θέμα αυτό και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα καταλήξει ε, η κατάσταση αυτή αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια γραμμή με την οποία συμφωνεί η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Στις 21 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, η ώρα 12. 16-17 Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή η ε, γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γεωργίας το Φεβρουάριο και μάλλον Μάρτιο-Απρίλιο θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και έτσι κλείσαμε και το σημείο 14 και πάμε πίσω στο σημείο 13. Εδώ Πρόκειται για τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την άσκηση των δραστηριοτήτων φάρμακοεπαγρύπνησης. Η Λίντα Μακάβαν είναι η συγγήτρια, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο. Ορίστε Λίντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξέρουν οι συνάδελφοι ότι είναι η τρίτη φορά που η Επιτροπή μας ασχολείται με την νομοθεσία όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση. Είχαμε για την ασφάλεια των φαρμάκων, τον έλεγχο των παρενεργειών, πώς ε, γίνεται η ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς αντιδράμε αν κάτι πάει στραβά. Κατά το παρελθόν είχαμε διάφορες περιπτώσεις, είχαμε το Mediator, το σκάνδαλο αυτό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μέσω νομοθεσίας που συμφωνήσαμε πρόσφατα Τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα νέο σύστημα φάρμακο Όταν πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε με αυτό και συμφωνήσαμε με αυτό, συμφωνήσαμε επίσης ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να πληρώνεται από τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις. Άρχισε να ισχύει νομοθεσία πέρυσι. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα συλλογής τελών, άρα πρέπει να εγκαθρεί αυτό το σύστημα, να δημιουργηθεί. Περί αυτού πρόκειται εδώ, σε αυτήν την ε, νομοθεσία. Το γεγονό ότι δεν υπάρχουν τέλη δημιουργεί προβλήματα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που είναι στο Λονδίνο και που έχει αναλάβει νέα καθήκοντα και αρμοδιότητε, αλλά δημιουργεί προβλήματα και στι χώρε μέλη, οι οποίες βασίζουν πολύ από τη δουλειά του. Βλέπετε, είναι ένας από τους οργανισμούς στον οποίο αποθύνονται οι χώρες ε, μέλη όταν έχουν γίνει μελέτες και τα λοιπά. Όταν όμως δεν χρηματοδοτούνται οι μελέτες αυτές δεν υπάρχουν. Συνεπώς το σύστημα που προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης αυτού του επιπλέον έργου το οποίο αποφασίσαμε να αναθέσουμε. Η συζήτηση λοιπόν είναι Ποιο πρέπει να είναι το ποσό των τελών αυτών, πώς θα προσδιορίζεται και όταν καθοριστεί το τέλος αυτό, πώς θα κατανέμεται ε, το ποσό που θα συγκεντρώνεται στις διάφορες ε, υπηρεσίες των χωρών μελών, στους εθνικούς οργανισμούς δηλαδή φαρμάκων. Τα τέλη τα χωρίζει η Επιτροπή σε δύο είδη. Το ένα είναι το καταποκοπήν τέλος, όπου θα πληρώνεται από όλε τι φαρμακευτικέ βιομηχανίε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το επιπλέον έργο που κάνει όσον αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση. Και το δεύτερο τμήμα του τέλου αυτού έχει να κάνει με συγκεκριμένα θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης και το ποσό κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ας έρθουμε πρώτα στο καταποκοπή. Ήδη παίρνει τέλη ο ΕΟΦ από φαρμακευτικές βιομηχανίες για διαδοτημένα προϊόντα. Παίρνει το λογαριασμό δηλαδή κάθε επιχείρηση γι' αυτό. Μετά όμως υπάρχουν και τα αποκεντρωμένα προϊόντα. Η δουλειά φαρμακοεπαγρύπνησης έχει να κάνει με προϊόντα όχι μόνο που είναι εγκριμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και επιμέρους. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ είχε μια ιδέα για το πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό το καταποκοπήν τέλος. Λένε ότι το συνολικό τέλος είναι κάπου 38 εκατομμύρια ευρώ. Το μισό ποσό θέλουν να είναι καταποκοπήν. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν το καταποκοπήν να βασίζεται στον αριθμό εισόδων στη βάση δεδομένων, τη Udra Vigilance. Βλέπω εδώ ότι ο κύριος κόλινς μου κάνει νοήματα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι βασιζόμαστε σε αυτόν τον αριθμό εισόδων στην βάση αυτή δεδομένων, το Udra Vigilance. Έχω κάποια προβλήματα όμως με αυτήν την ε, ιδέα του τέλους. Το πρώτο πρόβλημα που βλέπω είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι ο αριθμός ε, ημερησίων εισόδων είναι ο καλύτερος τρόπος για να καθοριστεί το τέλος. Γιατί κάποιοι μπορεί να κάνουν πολλές εισόδους. Κάποιος θέλει να δει για την συσκευασία, γιατί μπορεί να έχει ε, διαφορετικές συσκευασίες μια εταιρεία για το ίδιο της φάρμακο. Οπότε αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και έτσι προτείνω, αντί για αυτό, γιατί συζήτησα για το εφικτό της μεθόδου αυτής, προτείνω λοιπόν το τέλος που επιβάλλεται στην βιομηχανία, στην κάθε επιχείρηση, να εξαρτάται από τον αριθμό των αδειών που έχουν αδειοδοτηθεί. Τα δραστικά συστατικά δηλαδή. Να είναι ο αριθμός ε, αδειών που διαθέτει η εταιρεία αναδραστικό συστατικό. Το άλλο τώρα, έχοντας μιλήσει με τον ΕΟΦ για το επιπλέον έργο που αναλαμβάνουν, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως να μην εκτιμάει σωστά τα πράγματα. Μιλάτε για 90 εκατομμύρια ευρώ. Αν δείτε αυτό που προτείνω εγώ, αν αυξηθεί το ποσό ανά υποκείμενη σε τέλη μονάδα, τελικά μειώνεται το ποσό, γιατί θα υπάρχουν λιγότερα αδιαδοτούμενα προϊόντα τελικά. Να πω ότι τα δραστικά συστατικά. Νομίζω ότι 10,5 εκατομμύρια ευρώ θα συγκεντρώσουμε, που η Όφη λέει ότι είναι επαρκές ποσό για να καλυφθεί το επιπλέον κόστος που επομίζονται εκείνοι. Ορισμένε επιχειρήσεις ήδη πληρώνουν τέλη, οπότε δεν μπορούμε να επιβάλλουμε διπλό τέλος στις επιχειρήσεις αυτές. Προτείνω λοιπόν μείωση από αυτή την κεντρική διάθεση τελών και θέλω και τα σχόλια της Επιτροπής. Το άλλο είναι το θέμα των διαδικασιών. Όταν μπαίνει ένα φάρμακο στην αγορά. Αυτό δεν φτάνει. Οι επιχειρήσεις πρέπει να το παρακολουθούν, να το ελέγχουν. Γίνονται λοιπόν ε, εκθέσεις περιοδικές, ε, μελέτες ασφάλειας. Αν ένα φάρμακο παραπανθεί στον ΕΟΦ, τότε πρέπει να γίνεται μια διαδικασία κατεπήγοντος. Για αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα τέλος για τις φαρμακευτικές εταιρείες ως συμπληρωματικό τέλος. Οι επιχειρήσεις βέβαια μπορεί να κάνουν λόμπινγκ και να έρχονται και να σας λένε «Μα γιατί να πρέπει να πληρώσουμε κάτι παραπάνω». Μα η παραπάνω δουλειά που αναλαμβάνουν μειώνεται με την τελευταία διαδικασία. Για παράδειγμα, οι περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις ασφάλεια γίνονται από κάθε υπηρεσία, γινόντουσαν μάλλον από κάθε υπηρεσία, τώρα γίνεται μία ε, στον ΕΟΦ. για τις περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις ασφάλειας. Ωραία, προτείνει κάποιο τέλος που να κατανέμεται, επιτροπή μάλλον που προτείνει να κατανέμεται ανάμεσα στον ΕΟΦ και τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό το δέχονται όλοι. Το πρόβλημα έχει να κάνει όμως με την έκτακτη διαδικασία, την κατεπίγουσα. Όταν πρέπει να γίνει κάποια έρευνα από τον ΕΟΦ. Προτείνει κατά αποκοπή 168.000 που να πληρώνεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία και μπορεί να είναι πολλές επιχειρήσεις εξαρτάται πόσες είναι μαζί. Αν υπάρχει πρόβλημα με ένα φάρμακο, μπορεί να είναι τα δραστικά συστατικά, τα οποία να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά προϊόντα. Οπότε να είναι πολλές επιχειρήσεις μαζί που θα πληρώνουν το τέλος αυτό. Πάντως προτείνει κατά αποκοπή τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από ό,τι έχω καταλάβει, το εξηγήσει καλύτερη Επιτροπή, προτείνει 70% ΟΕΟΦ ή 25% για τα κράτη-μέλη, τέλο πάντων, κάπως έτσι, μια τέτοια κατανομή. Εγώ μίλησα και με το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη όμως από ό,τι φαίνεται κάνουν το μεγαλύτερο μέρο τη δουλειά για τις παραπομπές, όχι off. Οπότε τα κράτη-μέλη λένε αφού εμείς κάνουμε τη δουλειά γιατί να πάει το μεγαλύτερο ποσό off. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο Συμβούλιο επί του παρόντο. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σχολιάσει. Δεν προβαίνουν σε αλλαγέ. Δεν κάνω για να αλλάξω την ισορροπία ανάμεσα στον ΕΟΦ και τα κράτη-μέλη. Παρόλο που σας λέω στο Συμβούλιο, είναι πρόβλημα. Ο εισηγητής ορίζεται από ένα κράτος μέλος και ορίζονται και συνεισηγητές για να δουλέψουν πάνω στην ίδια παραπομπή. Αυτό κοστίζει χρήματα. Και τα κράτη-μέλη λένε ότι τους κοστίζει και πολύ χρόνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή προτείνει το καταποκοπή τέλος 168.000, αλλά δεν είναι πάντα όλες οι παραπομπές εξίσου περίπλοκες. Γι' αυτό εγώ προτείνω να μην έχουμε καταποκοπή ποσό για τις παραπομπές, αλλά διαβαθμισμένο. Να λέμε ότι μία παραπομπή μπορεί να χρειάζεται 5, 6, να φέρει σε 5-6 δραστικέ ουσίε, μια άλλη σε μη δραστική ουσία. Οπότε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Συμφωνεί το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο ΟΦ να αποφασίζει για το τέλο ανάλογα με τη δουλειά που χρειάζεται στην περίπτωση τη κάθε παραπομπής. Πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο τέλο και τη δουλειά που γίνεται, γιατί μετά θα έρθει το ελεγκτικό συνέδριο και θα πει μα Οπότε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σχολιάσει αυτό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ορισμένες κατηγορίες να αποκλειστούν από την πληρωμή τελών γενικά. Μιλάμε εδώ πώς τα λένε, έχω χάσει εδώ τα χαρτιά μου, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Προτείνουν λοιπόν τα κατοχωρημένα ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά να μην συμπεριληφθούν στην νομοθεσία. Έχω δεχτεί πολλοί λόμπι από διάφορες επιχειρήσεις. Σας μας το διευκρινίσει αυτό για τα καταχωρημένα βοτανοθεραπευτικά και ομοιοπαθητικά φάρμακα κατά πόσο θα αποκλείονται από τα τέλη, θα εξαιρούνται από τα τέλη, όπως και κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα ισχύει το ίδιο. Όμως για αυτά που έχουν άδεια, γιατί τα γενώσιμα και τα... αυτά που έχουν άδεια καθιερωμένης χρήσης δεν νομίζω ότι παίρνουν εξαίρεση. Για τα γενώσιμα θέλω να ρωτήσω όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εσείς προτείνετε μια μείωση. Όταν ρώτησα τον ΕΟΦ, που έχουν 20% βάσει της πρότασής σας μείωση, σε συνδυασμό με αυτό που προτείνω για την αλλαγή στο καταποκοπή ποσό να μην είναι πια καταποκοπή, οπότε δεν θα πληρώνουν ένα πακέτο καθημερινά, αλλά ανάλογα με τα δραστικά συστατικά, άρα κερδίζουν από αυτό. Οπότε όταν ρώτησα τον ΕΟΦ για τον αριθμό παραπομπών που έρχονται για τα γενώσιμα, μου είπαν ότι μισές παραπομπές, περισσότερες από τις μισές παραπομπές το 2009 μέχρι το 2013 ήρθαν από επιχειρήσεις γενώσιμων φαρμάκων. Τώρα το ότι είναι γεννόσιμα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή, οπότε χρειάζονται παραπομπές. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί να τους δίνουμε μείωση στις παραπομπές εφόσον αυτά τα γεννόσιμα είναι ακριβώς αυτά που είναι η αιτία για τον μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών. Θέλω να καταλάβω και τη διαφορά ε, της καθιερωμένης χρήσης. Είναι επιχείρηση που το επιλέγει αυτό. Σε ορισμένες χώρες κάποια γενώσιμα θεωρούνται καθιερωμένες χρήσεις, αλλά όχι, θέλω να μου το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να καταλάβουμε δηλαδή τον αριθμό τελών που συγκεντρώνουμε. Τέλος πάντων πρέπει να υπάρξει σύντομα συμφωνία γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια νομοθεσία για μια δουλειά που γίνεται και που δεν αμείβεται. Δύο χρόνια χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει την πρότασή της και τώρα εμείς πρέπει να βιαστούμε πριν τις εκλογές. Στο Συμβούλιο, από ό,τι καταλαβαίνω, επίσης επιταχύνονται τα πράγματα. Πάντως, η πιο πρόσφατη θέση στο Συμβούλιο είναι ότι το Συμβούλιο θέλει να διαγράψει τα κεντρικά τέλη για τον ΕΟΦ. Είναι το τελευταίο που άκουσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα από την ομάδα εργασία. Οπότε δεν χρηματοδοτείται έτσι η δουλειά του ΙΟΦ για την φαρμακοεπαγρύπνηση. μια Επιτροπή τι λέει, εμένα δεν μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό. Εγώ νομίζω και τα αποκεντρωμένα και τα άλλα πρέπει να υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εξαφανιστούν. είναι ουσιαστικά τα δύο σκέλη της ρυθμιστικής διαδικασίας που χρηματοδοτούμε. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου ή αμέσως μετά θα προτείνει και ένα τρίτο κανονισμό για τα τέλη φάρμακο επαγρύπνησης και για τη χρηματοδότηση του ΕΟΦ. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια γρήγορη λύση για να χρηματοδοτηθεί το έργο και αν θέλετε επαναστατικές αλλαγές μπορούν να περιμένουν να γίνουν μετά από δύο χρόνια που θα συζητήσουμε γενικά για τη χρηματοδότηση του ΙΟΦ. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Ξέρω ότι ορισμένοι χαίρονται για το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω. Αν πρόκειται να συμφωνήσουμε και θέλουμε να έχουμε χρόνο για τριμερή διάλογο κτλ. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι πάει τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Αν αργήσουμε περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Θέλω να καλωσορίσω κάποιον εδώ. Ο, ο δράστης γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, όπως ο Κιν Κόλλινς, ο προκάτοχός μου, ο οποίος φράγησε την Επιτροπή. Ε, ε λέει ότι τον θυμάται πολύ καλά από τα παλιά μέλη. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στους κόλπους μας. Και τώρα η Σκιώδης, η Πιλάρα Γιούζο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την κυρία Μακάβεν για την έκθεσή της και για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί της. Όντως πάμε πολύ καλά οι Σκιώδης μαζί της. Συμφωνώ λίγο πολύ με όλα όσα μας είπε. Συμφωνώ οι συγητές και οι συγητές από τις χώρες μέλη να αμείβονται για το έργο τους. Επίσης να υπολογιστούν τα τέλη ανάλογα με το δραστικό συστατικό και να λάβουμε υπόψη μας και το μέγεθος της συσκευασίας το γεγονός ότι υπάρχουν 60 μέρες για την πληρωμή των εισηγητών είναι και αυτό μια καλή πρόταση νομίζω. Τώρα για τα γενώσιμα φάρμακα. Δεν θα πρέπει να αποκλείονται. Ιδίως μάλιστα εφόσον προκαλούν επιπλέον δουλειά για τον ΕΟΦ. Πρέπει να συμμετέχουν στο τέλος, να πληρώνουν τέλος και αυτές. Όσον αφορά τώρα την αύξηση του ετησίου τέλους που προτείνει η συγκήτρια, πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το ποσό και τη το είπα και σε προηγούμενη συνάντησή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να μας διευκρινίσει ποιο είναι το κριτήριο που ακολουθεί για να υπολογίζει το ποσό αυτό. ιδίω αν λάβουμε υπόψη μα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε βάθος αναδιάρθρωση του συστήματος σε λίγα χρόνια. Για την αμοιβή λοιπόν εγώ θα ήθελα να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι αποκλειστικές αρμοδιότητες του ΕΟΦ για τις οποίες πρέπει να χρηματοδοτείτε και ποιες είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αυτό είναι κάτι πιστεύω σημαντικό, ιδίω όταν μιλάμε για χρηματοδότηση. Περιμένω λοιπόν τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις δικές μου ερωτήσεις αλλά και σε εκείνες της εισηγήτριας. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Αντώνια Παρβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον την εισηγήτρια. Όλοι της έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Φαίνεται αυτό από τη δουλειά της με τους Σκιώδης. Υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής συνεργασία και στον προηγούμενο γύρο του φακέλου φαρμακοεπαγρύπνησης παρά το γεγονός της καθυστέρησης από την Κομισιόν που δεν συγχώνευσε έγκαιρα τους δύο φακέλους, παρόλα αυτά μπορεί να προλάβουμε και να κλείσουμε το θέμα στη θητεία του Κοινοβουλίου. Θα πιεστεί λίγο το Συμβούλιο. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις από πριν. Πάντως, θέλω να πω ότι το βασικό θέμα είναι η απλότητα και η διαφάνεια. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα υπήρξαν κάποιες εντάσεις και συγκρούσεις απόψεων για το αν ο ΕΟΦ θα έπρεπε να παίρνει κι άλλα τέλη από το κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και αν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Αλλά επειδή αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει και υπάρχουν παρόμοιες πρακτικές κι αλλού, δεν είναι κακό να πληρώνει κανείς για τις υπηρεσίες που παρέχονται, ούτε υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και βεβαίως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου ΕΟΦ θα πρέπει να χρηματοδοτείται καλά όχι μόνο από τον προϋπολογισμό, αλλά και από αυτούς που τον χρησιμοποιούν. Τώρα για τις ε, δραστικές ουσίες συμφωνώ με την εισηγήτρια για να μην ε, ε, υπάρξουν δυσκολίες αν στηριχθούμε στο μέγεθος της συσκευασίας. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η ίδια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί και για τα γενώσιμα. Εγώ προτιμώ να υπάρχει ετήσιο καταποκοπήν ποσό, γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κράτη-μέλη το μέγεθος συσκευασία. Γιατί για ιστορικούς λόγους εκεί απαιτείται πιο πολύ και λεπτομερής διαχείριση. Πάντω μπορούμε ε, από κοινού να διευκρινίσουμε τα θέματα αυτά και ε, θα πρέπει και η Κομισιό να μας πει τι εκτιμήσεις κάνει, αν κάνει σχετικά με τον αντίκτυπο που θα υπάρξει από τη μία ή την άλλη προσέγγιση. Και γενικά περιμένω με χαρά να συνεχίσω τη συνεργασία μου την κυρία Μακάβαν και σίγουρα θα έχουμε μεγάλη επιτυχία και ένα πολύ καλό φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Γιανακουδάκη Μαρίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Λίντα για την εργασία της μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι ε, σαν μπούμεραγκ αυτό το θέμα, σαν κακό όνειρο. Ε, σας ξαναβρίσκει κάθε φορά και έχουμε φτάσει τώρα στο τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου. Ε, ανησύχησα πάρα πολύ όταν μας ζητήθηκε μια τόσο γρήγορη έκθεση. Ε, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν συμφωνεί με κανέναν άλλον. Ε, υπάρχουν 7-8 διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ε, ένα πράγμα που με ανησυχεί είναι συνολικά η ιδέα αυτού του θέματος για το κατά πόσον χρειαζόμαστε αυτά τα τέλη. αλλά τελικά δεν είμαι σίγουρη εφόσον σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε μια ε, πλήρη αλλαγή της νομοθεσίας γιατί χρειάζεται να παραγάγουμε κάτι τόσο γρήγορα, ε, τόσο βιαστικά. Υπάρχουν και άλλα σημεία που με ανησυχούν όσον αφορά τα τέλη. Θα ήθελα να είναι αναλογικά και νομίζω ότι η Κομισιόν εδώ έχει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση από την ε, αίμα, από ό,τι ανακαλύψε η Λίντα. Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται διπλά τέλη. Το όλο σύστημα βασίζεται σε ένα σύστημα μηχανοργάνωσης ε, του αίμα που δεν φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και αυτό θα προκαλέσει προβλήματα. Ε, υποστηρίζω τη Λίντα σε αυτό που λέει για την προσέγγιση βάση των ε, δραστικών ουσιών, αυτά που λέει για τα γενώσιμα και για τα βοτανοθεραπευτικά φάρμακα και τα μεβοθητικά. Κάτι που με ανησυχεί είναι ότι ε, εξουδοτούμε την Κομισιόν να χρεώσει κάποια τέλη ε, από μόνη της αργότερα. Θα πρέπει να έχουμε έλεγχο πάνω σε αυτό. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι η συγκήτρια θα καταλήξει σε μια πολύ καλή έκθεση με την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ η κυρία Σούζα για το Ιγκούε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατη. Πολλές πτυχές αυτής της έκθεσης νομίζω ότι χρειάζονται διευκρίνηση. Ήδη ζήτησε διευκρινήσεις η εισηγήτρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να συγχαρώ τη Λίντα για την εργασία της μέχρι τώρα. Θα είναι δύσκολο το έργο μας. Μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι και τα εξή. Η κυρία Μακέβαν βελτίωσε κατά πολύ την πρόταση της Κομισιόν, οπότε αυτό είναι καλό σημείο εκκινήσεως, αλλά όπως είπε και η ίδια, ακόμα χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις από την Κομισιόν Ιδάλος. Θα έχουμε πρόβλημα κι εμείς η σκιωδηση γιατί δεν θα καταλαβαίνουμε ακριβώς τι προτείνει η Κομισιόν. Θέλουμε να αποφύγουμε τη διπλή χρέωση και εις ό,τι αφορά τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, Ίσως θα έπρεπε να τους δίνουμε πιο πολύ χρόνο για να πληρώνουν τα τέλη, ιδιαίτερα σε χώρες με οικονομικό πρόβλημα, συνεχιζόμενο και επιδεινούμενο. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε σε τέτοιου είδους ε, χώρες μέλη και άλλα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και δυσκολίες. Και οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις τώρα έχουν ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να πληρώσουν. Και έτσι μπορεί να μην προλαβαίνουν να παράγουν τα φάρμακα και να τα βγάζουν στην αγορά. Σταματώ εδώ, έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε περισσότερο, θα είναι μια δουλειά ε, πολύ καρποφόρα, αν και βεβαίως ε, οι προθεσμίες είναι πολύ περιορισμένες και πιεστικές και δεν ξέρω πώς οι προτάσεις αυτές θα συνάδουν και με τις ε, μελλοντικέ και γενικότερες προτάσεις που θα υποβάλει σε εμάς η Κομισιόν. Σε εμάς όταν λέω όχι σε αυτή τη θητεία. Και αυτό είναι μια αντίφαση, γιατί εμείς κάνουμε δουλειά για τμήμα ενός συνόλου, το οποίο σύνολο θα διακοπεί κάποια στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε τι συνέχεια θα δοθεί και πώς θα ενταχθεί στο γενικότερο προγραμματισμό. Ευχαριστώ. Και τώρα η Dagmar Ροτμπέρεν που είναι ο σύνδεσμος με τον ΕΟΦ τεχνικό πρόβλημα. Δεν κάνω παρεμβολές, εγώ δεν έχω το κινητό μου κοντά, δεν φταίω για τους ήχους που ακούμε. Α, ο Κέν έφταιγε. Όχι, ούτε ο Κέν έφταιγε. Α, εδώ, εδώ, εδώ. It does not Sind unterwegs? Λοιπόν, στείλαμε να φωνάξουμε τους τεχνικούς. Είναι καθοδόν, έρχονται. Τώρα εδώ, εδώ είναι καλύτερα. Μου φαίνεται, τι είναι αυτό. Κάποιος ήθελε να με χωρίσει από τον Κεν. Λοιπόν, δύσκολη πρόταση, καθυστερημένη, όψιμη και κοιτάζω την Κομισιόν εδώ. Θα μπορούσαν να μας την υποβάλουν πολύ νωρίτερα. Τώρα μας βάζουν να τρέχουμε. Εσείς φταίτε που τρέχουμε τώρα. Γιατί η πρώτη πρόταση ήταν εξωφρενική. Και μέχρι τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν έφταιγε η Κομισιόν, αν έφταιγε ο ΕΟΦ. Τέλος πάντων δεν με απασχολεί αυτό. Τώρα έχουμε μία πρόταση που είναι προώρη για να το θέσω ήπια. Κάποια στοιχεία είναι κατανόητα, αλλά και δεν βλέπω συνοχή στην όλη προσέγγιση. Ελπίζω η έκθεση της Λίντα Μακάβαν και οι τροπολογίες μας να την φτιάξουν λίγο και να την κάνουν να έχει περισσότερη συνοχή. Για να δούμε τα επιμέρους. Όταν μιλάμε για φαρμακοεπαγρύπνηση, μιλάμε για πιθανό κίνδυνο, έτσι, ενδεχόμενο κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Σήματα που θα έρθουν από τα φαρμακευτικά προϊόντα. Έτσι τα ομοιοπαθητικά και κάποια άλλα αποκλείονται αυτομάτως. Το είπες εσύ πολύ σωστά Λίντα. Όταν μιλάμε για προϊόντα όπως ας πούμε βότανα με εδρεωμένη δράση και χρήση είναι σαφές ότι η πιθανότητα να υπάρξει κάποιο σήμα κινδύνου είναι σχεδόν μηδέν, μηδενική. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη σε κάθε κομμάτι της νομοθεσίας και δεν το έχετε κάνει όπως έπρεπε. Όταν μιλάμε για φαρμακοεπαγρύπνηση και θέματα δημόσιας υγείας, αναρωτιέμαι γιατί η πρόταση δεν αναφέρει πουθενά ότι εδώ πρόκειται για θέμα δημόσιας υγείας. Δηλαδή τις δημόσιες αρχές δεν τις λαμβάνει υπόψη καθόλου. Και τι ευθύνες έχουν αυτές. Η ό,τι αφορά τις ε, ευθύνες και τις αρμοδιότητες, αυτό είναι λάθος. Επίσης είναι λάθος ε, διότι συμπεριλαμβάνουμε και εθνικές διαδικασίες ε, αδειοδότησης ή εξουσιοδότησης. Αν πείτε ότι είναι συγκεντρωτικό και ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργεί το συγκεντρωτικό σύστημα και να είναι καλό. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό διαδικασιών εξουσιοδότησης ή έγκρισης εθνικών, από εθνικές αρχές. Μπορεί να πάρουν καλά τα πράγματα εκεί, μπορεί και όχι. Και αναφερόμαστε όλο και περισσότερο σε παλαιότερα προϊόντα και γενώσιμα. Γι' αυτό η μείωση για τα γενώσιμα είναι γελία πρόταση. Γιατί είναι σαφές ότι όσο πιο παλιό είναι ένα προϊόν, και αυτό λέει και ο ΕΟΦ, τόσο περισσότερα μηνύματα θα έρχονται γι' αυτό και σήματα. Είναι πολύ πιο πιθανό το παλαιότερο να είναι γενώσιμο γιατί μπορεί να έχει ε, λήξει και η άδεια ευρεσιτεχνίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα γενώσιμα που είναι αντίγραφα ενός χημικού προϊόντος μπορεί να έχουν παρόμοιες ανιχνεύσεις ενδείξεων. Γιατί λοιπόν να υπάρχει μείωση των τελών για τα γενώσιμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πάμε σε άλλες ε, εκπτώσεις, μειώσεις τελών. Έχετε για σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες. Ανέφερε και η ε, κυρία Σούσα αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που αλλά ε, ο ορισμός ε, των ΜΜΕ της Κομισιόν είναι περίεργος. Αν θέλει να αναφερθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μιλήσει για πολύ μικρές επιχειρήσεις, για πολύ μικρά εργαστήρια ή για την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται. Αλλά όχι να ε, φέρνετε εδώ ένα τέτοιο ορισμό όπως αυτόν που έχετε εδώ. Ο ύστερα, πώς το σύστημα. Νομίζω ότι το ετήσιο τέλος καλή ιδέα είναι. Αλλά το ετήσιο καταποκοπή που είναι είναι μόνο καλή ιδέα, εκεί στο άρθρο 7, αν υπάρχει σωστός ορισμός της χρεώσιμης μονάδας. Και τώρα το έχει αλλάξει η Λίντα. Εσείς δεν το κάνατε, γιατί δεν την εξετάσατε αυτή την ιδέα, ότι ξαφνικά μπορεί να υπάρξουν τεράστιοι αριθμοί ε, που θα αφορούν προϊόντα απλά σε μεγάλη όμως συσκευασία. Αν θέλουμε να δούμε το ετήσιο κατά αποκοπήν ποσό, τέλος πρέπει να έχουμε τη χρεώσιμη μονάδα, σωστό ορισμό, πρέπει να αλλάξει, να δούμε τις δραστηριότητες που πρέπει να διευκρινιστούν από, την, ε, από τον ΕΟΦ και να προσαρμόσουμε ανάλογα το ποσό και να έχουμε σαφείς τρόπους ε, για το ε, λειτουργία του συστήματος διακρίσεων και μειώσεων. Για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το ποιος θα κάνει τη δουλειά. Το είπα και χθες όταν ε, συζητούσαμε με τον ΕΟΦ. Κάποιοι δεν μπορέσατε να έρθετε. Ο Γκουίντο Ράζι όμως είχε έρθει εδώ. Και κάναμε καλή συζήτηση. Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου είπε και ο εκπρόσωπος του, του Κοινοβουλίου είναι ότι θέλουμε να έχουμε στην νομοθεσία λόγο. Εγώ ελπίζω να ήμουν αρκετά ευγενική και σαφής όταν είπα ότι είναι συνομοθέτης με το Συμβούλιο του Κοινοβούλιο και σε κάποιο στάδιο η Κομισιόν. Όχι όμως το Διοικητικό Συμβούλιο της του ΕΟΦ που δεν πρέπει να έχει λόγο. Και ε, όταν θέλουμε να κάνουμε τροποποίηση της νομοθεσίας. Η συνάδελφος Γιάννα Κουδάκη μίλησε για εντεταλμένες αρχές, ε, φαντάζομαι μιλούσες για εξουσιοδοτημένες πράξεις. Συμφωνώ, καλό πράγμα είναι να χρησιμοποιήσουμε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει αντίρρηση και κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Αλλά αν θέλετε να πάτε μέσα από κατεξουσιοδότηση πράξης, αυτό θα γίνει μόνο ε, με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου. Και επειδή στο παρελθόν πολλές φορές αποτύχατε να χρησιμοποιήσετε τις κατεξουσιοδότηση, θα πρέπει να το σκεφτείτε. Καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι. Τώρα, με τις παραπομπές τι θα κάνουμε. Το τέλος παραπομπής, 160.000 ευρώ για την παραπομπή, όπως ξέρουμε όλοι, αυτό ε, είναι, έχει εφευρεθεί. Να φέρετο. Πήρατε χιλιάδες ώρες παρουσίας από εθνικό οργανισμό, ενώ ξέρουμε ότι αυτό είναι αυθαίρετο και δεν ε, είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ορισμένα πράγματα εδώ. Πρώτον, ναι, υπάρχουν χρήσιμες παραπομπές. Υπάρχουν όμως και άσκοπες παραπομπές και όταν μια εθνική, και συμβαίνουν όταν θέλει να απεκδηθεί των ευθυνών της η εθνική αρχή. Πρέπει λοιπόν να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ, εδώ και πάλι, μεταξύ εθνικής διαδικασίας και ε, συγκεντρωτικής διαδικασίας αδειοδότησης. Η Εθνική Αρχή έχει μεγάλες ευθύνες για την έγκριση ε, στο κράτος μέλος. Υπάρχει βέβαια και η αμοιβαία αναγνώριση για να ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη. Τώρα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος. Πρέπει. Γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας αυτό. Παράλληλα πιστεύω ότι κάθε εθνική αρχή που φέρνει μια παραπομπή στον ΕΟΦ δεν μπορεί να είναι ούτε συγητής ούτε Διότι αυτό θα ήταν μια σύγκρουση συμφερόντων ε, μία αντίφαση απαράδεκτη. Τώρα και πάλι, ποιος, λέμε, ποιος κάνει τη δουλειά. Μπορούμε να πούμε ότι θα τα κάνει όλα μόνη της ο ΕΟΦ, μόνος του ΕΟΦ. Δεν θα με εμένα αν λέγαμε παράλληλα ότι τα κράτη-μέλη και οι εθνικές αρχές των κρατών μελών έχουν λόγο και μπορούν να είναι εισηγητές και θα πρέπει να αμείβονται για τη δουλειά τους. Τότε συμφωνώ να το κάνουμε έτσι, αλλά θα πρέπει τότε να ξέρω γιατί θα παίρνουν τα λεφτά. Και πρέπει να, είμαι πολύ σαφ... πρέπει να είναι πολύ σαφές πόσες ώρες θα δουλεύουν πάνω σε τι. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ε, λεπτομερές ωράριο και περιεχόμενο εργασίας. Οι εθνικές αρχές μπορεί να πούνε βέβαια ότι ούτε ο ΕΟΦ το κάνει αυτό. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Είναι δημόσια αρχή ο ΕΟΦ που αναθέτει καθήκοντα σε άλλους. Θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ο ΕΟΦ θα τα κάνει όλα. Δεν θα με νοιάζει. Στο βαθμό όμως που θέλουν να συμμετέχουν στη δουλειά οι εθνικές αρχές που είναι καλό τότε θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν μερίδιο σε όλα αυτά. Ε, τώρα πώς θα ορίσουμε τα ποσά. Η Λίντα είπε και το, έβγαλε το ποσό από την πρόταση. Είπε πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούμε πάλι αυτό και να δούμε πώς θα χειριζόμεθα τις παραπομπές. Γιατί μια παραπομπή μπορεί να επηρεάζει γιατί ένα προϊόν μπορεί να παραπενθεί και αυτό ναι, έχει αντίκτυπο σε χιλιάδες, σε χίλια, δύο χιλιάδες άλλα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε προσεκτικά. Τέλος, πρέπει να προσέξουμε πολύ, να τα κάνουμε σωστά. Τα μέτρα λιτότητας ε, όπως μας εξήγησαν τα κράτη-μέλη, σημαίνει ότι ε, μειώνονται τα χρήματα για τις δημόσιες αρχές. Πρέπει να ε, ε, τρέχουν στον ενωσιακό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι σωστό αυτό, υπάρχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτή την πρακτική για πολύ καιρό, υπερβολικά πολύ καιρό τη δεχτήκαμε. Τώρα γίνονται άπληστοι, όπως βλέπουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, υπό την ηγεσία κανένα δύο κρατών μελών, δεν ξέρω και το δικό μου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλουμε να έχουμε σαφέστατο ορισμό σχετικά με το κόστος παραπομπής, ποιο είναι, τι θα πληρώνετε από το δημόσιο να το πω. Να το πω. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Τι πληρώνουν οι διάφορες εταιρείες, τι πληρώνουν στους εισηγητές και συνεισηγητές και βέβαια δεν θα πρέπει η αρχή που κάνει την παραπομπή να είναι εισηγητή ή συνεισηγητή. Για το καταποκοπήν η Λίντα έχει δίκιο, πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι καλύπτει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε ότι θα είναι ξεκάθαρο ότι ο ΕΟΦ θα πρέπει να ψάξει την, την βιβλιογραφία και ενδελεχώς μάλιστα να κάνει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφία γιατί δεν υποχρεούνται οι εταιρείε, γιατί με το καταποκοπήν ποσό θα καλυφθούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που ίσως ποτέ δεν θα στείλουν ε, μήνυμα ή θα κάνουν ανείχνευση ενδείξεων και όταν θα πρέπει να έχουμε κατά αποκοπήν ποσό και όταν το πληρώνουν πρέπει να παίρνουν και κάποιες υπηρεσίες που θα αναλογούν στα λεφτά που θα πληρώνουν. Να το φροντίσουμε αυτό. Ε, υπάρχει περιθώριο να καταθέσω τροπολογίες. Ελπίζω μέχρι την Παρασκευή, προλαβαίνω δεν προλαβαίνω, θα κοιτάξω να τα καταφέρω. Ας πάει όμως την προθεσμία Παρασκευή βράδυ. Έτσι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ε, ζητώ συγγνώμη που το ζητώ αυτό, ξέρω πόσο σκληρά δουλεύετε, αλλά αν πάει η προθεσμία κατάθεσης ε, Παρασκευή βράδυ θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Καλώς. Και η Κομισιόν τώρα παρακαλώ. Ποιος θέλει πρώτος, ο κύριος Ρης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια και τους ε, σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους. Χαίρομαι που παρατηρώ ότι ε, όσον αφορά την ουσία ε, της πρότασης αυτής δεν προβλέπεται να έχουμε ουσιαστικές δυσκολίες εκ μέρους της Κομισιόν. Αλλά για τις τροπολογίες 3, 9, 12, 14 θα αναφερθώ σε αυτές και θα απαντήσω και σε μερικές συγκεκριμένε ε, ερωτήσεις. Όσον αφορά την έκπτωση για τα γενώσιμα, ε, στην πρότασή μας θεωρούμε ότι η μείωση των τελών για τα γενώσιμα δεν δημιουργεί ασυνέπεια προτείνουμε μείωση 20% όσον αφορά το ετήσιο καταποκοπή τέλος για τα γενώσιμα ή για φάρμακα που έχουν ε, άδεια καθημερινής χρήσης ή για βοτανοθερπευτικά και ομευτικά με άδεια κυκλοφορίας. Έγινε μια ερώτηση σχετικά με το ποιο, πόσο ορίζονται τα γενώσιμα ή τα φάρμακα με άδεια καθημερινής χρήσης αυτό είναι συνεπές με την νομοθεσία για την φάρμακοεπαγρύπνηση που εξαιρεί ε, τα προϊόντα αυτά από την υποχρέωση ε, υποβολής περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για την ασφάλεια γιατί τα προϊόντα αυτά θεωρούν ότι έχουν καθιερωμένο προφίλ ασφαλείας, ε, εδρεωμένο. Τα γενώσιμα ανήκουν στην κεντρική διαδικασία και σήμερα ήδη αποφελούνται από πολύ σημαντικές ε, εκπτώσεις. 70% από το ετήσιο τέλος που ισχύει για, τα, ε, για την έγκριση προϊόντων. Άρα είναι συνεπές κατά τη γνώμη μας αν ε, σε εθνικό επίπεδο δεν θα υπάρχει καμία μείωση. Όμως η έκπτωση που προτείνεται για τα γενώσιμα βασίζεται σε καλά εδρεωμένο ε, προφίλ ασφαλείας ε, σε σχέση με τα άλλα προϊόντα. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει μείωση για τα ε, έξοδα, για τα τέλη διαδικασίας παρά μόνο για το καταποκοπή τέλος. Όσον αφορά την τροπολογία 13 ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης εδώ, ε, εμείς θα προτιμούσαμε να ορίζουμε κάποια ποσά και όχι ποσοστά σε ένα νομικό κείμενο. Η πρότασή μας βασίζεται σε μια εκτίμηση ενός μέσου κόστους για το αίμα και για τους συγητές από τα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι με βάση αυτή την προσέγγιση είναι προτιμότερο να αναφερόμαστε σε συνολικό ποσό και όχι σε ποσοστό για να δείξουμε ότι η πρότασή μας βασίζεται στο κόστος. Προσπαθήσαμε να πάρουμε όλα τα στοιχεία που είχε ο ΕΜΑ και τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε στην ε, οριστική μας πρόταση. Συλλέξαμε πάρα πολλά τέτοια επίσημα στοιχεία. Όσον αφορά το ποσό που αναφέρεται στην τροπολογία 14, ε, η αύξηση από 60 σε 168.000 ε, για το καταποκοπή τέλος, αυτό σχετίζεται με την χρεώσιμη ομάδα. Ε, γι' αυτό υπάρχει υψηλότερο αιτήσιο κατά αποκοπή τέλος. Και θα θέλαμε εδώ να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν διάφορες μεταβλητές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ιδιαίτερα ε, ο αριθμός των χρεώσιμων μονάδων που δεν θα παραμένει σταθερός. Γι' αυτό ε, υπάρχει ανάγκη ε, ευελιξίας για την Κομισιόν ώστε να μπορεί να προσαρμόζει ε, αυτό το ποσό αν χρειαστεί. Και χαιρόμαστε που τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αρχίσαμε να υπολογίζουμε τον αριθμό των προϊόντων για την πρόταση που κάνουμε, μιλούσαμε για περίπου μισό εκατομμύριο προϊόντα Σύμφωνα με την πρόταση της εισηγήτριας θα είναι το ποσό αυτό, η ποσότητα αυτή 130.000. Ε, και το κόστος λόγω της αλλαγής του πεδίου εφαρμογή θα μειωθεί από 19 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια. Αυτό αντιστοιχεί στις προτινόμενες δραστηριότητες από την εισηγήτρια. Όσον αφορά όσον αφορά τις αμοιβέ και το χρονοδιάγραμμα για τους ηγητές ε, στην τροπολογία 12 για τις 12 μέρες από την παραλαβή της έκθεσης κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται να προβλέπετε μια προθεσμία ε, για τις αμοιβέ αυτές μέσα στον ίδιο τον κανονισμό ε, η αμοιβή για τα κράτη-μέλη είναι θέμα που θα πρέπει να ρυθμίσουν μεταξύ του τα κράτη-μέλη και ο αίμα, όπω και άλλοι κανόνε. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν ε, συμφωνίε συνεργασία μεταξύ ε, του αίμα και των αρμοδίων εθνικών αρχών. Αυτό είναι μια πιο εύκολη και πιο ευέλικτη λύση και πιο εύκολο να αλλάξει η ρυθμίση αυτή αν χρειαστεί. Ε, ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα σχετικά με το μοίρασμα του κόστους των εργασιών την κατανομή του κόστους. Είναι σαφές ότι μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του συστήματος ο ΕΜΑ έχει πολύ πιο ξεκάθαρες ιδέες για το πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιο είναι το κόστο. Παραδείγματο χάρη, ο ΕΜΑ αναφέρεται στο θέμα του ΠΡΑΚ ε, και άλλες δραστηριότητες αλλά και πάλι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε υπό το φως ε, της ε, πρότασης για να τα καθορίσουμε σωστά. Ε, στο Συμβούλιο συνεχίζεται επίσης η συζήτηση. Τα κράτη-μέλη έχουν δώσει πρόσθετα στοιχεία τις, τις τελευταίες εβδομάδες και ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπίας της κατανομής των ε, εργασιών και του κόστους ανάμεσα στον αίμα και στις εθνικές αρχές. Συμφωνούμε με την πρόταση σχετικά με τα ομοιοποθητικά και τα βοτοαναθεραπευτικά προϊόντα που θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτή την πρόταση όταν έχουν καταχωρηθεί. Ε, ναι, έχει νόημα να μπει αυτό μέσα στον ίδιο τον κανονισμό, συμφωνούμε. Όσον αφορά την κατάσταση στο Συμβούλιο, είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, του Συμβουλίου αμφισβητήθηκε το καταποκοπή τέλος ε, και το κατά πόσο ήταν αυτή η σωστή προσέγγιση. Όπως έχουν σήμερα όμως τα πράγματα, έχουν επανέλθει, έχουν αλλάξει γνώμη, άρα αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι αυτή η μεικτή προσέγγιση, δηλαδή η καταποκοπή τέλος, στην προσέγγιση ε, αναεπιφάνεια, ε, λειτουργεί καλύτερα. Επίσης είναι γεγονός ότι το όλο αυτό εγχείρημα είναι μια καλή στιγμή για τον αίμα και για τις εθνικές αρχές, αλλά και για μας ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσουμε τον ευρύτερο ε, κανονισμό για, για τα τέλη με βάση το πραγματικό κόστος. Θεωρούμε λοιπόν ότι με βάση την εξέλιξη όλων των εργασιών εδώ και στο Συμβούλιο ε, ότι υπάρχουν αρκετά δύσκολα ζητήματα ε, σχετικά με τα δεδομένα, σχετικά με το πώς βλέπουν το κόστος οι διάφορες εθνικές αρχές και η δομή των διαφόρων φορέων ε, ποικίλει από κράτος σε κράτος. Τέλος, ε, με χαρά μας θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μαζί σας και θα σας ε, παρέχουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με σκοπό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η, η συγγήτρια τώρα. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι ήθελε να απαλλαγεί από την ιδέα του κατά αλλά πρέπει να του θυμίσουμε ότι αν οι μετα ΜΜΑ, οι μεταναλύσεις αυτές με τα, τις μελέτες στοιχίζουν, ε, θα είναι και τα τέλη ψηλά. Γιατί θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα κόστη και επέμειναν, είπαν ότι δεν θα συμφωνούσαν. Και κατάλαβα ότι ε, θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Ε, Τώρα, εγώ δεν θέλω να επιβληθεί τέλος σε επιχειρήσεις. Το αντίθετο, αν αλλάξω με τον ορισμό της χρεώσιμης μονάδας, πάμε στα υδραστική, τότε το ποσό θα είναι το μισό. Δεν έχω τα στοιχεία από την Κομισιόν, αλλά ζήτησα κάποια στοιχεία για να δω πόσο πληρώνουν οι κατά μέσον όρο. Δεν μου απαντήσαν, αλλά πληρώνουν λιγότερα. Είναι λιγο, ε, θα, θα, πληρώνουν λιγότερο. Ε, δηλαδή το μπορεί να πληρώνουν λιγότερες φορές 86 σε σχέση με περισσότερες φορές 60. Ε, ο ΕΟΦ τώρα υπολογίζει, ο ΕΜΑ δηλαδή, ε, ότι μπορεί να αναλάβει κάποια καθήκοντα φάρμακο επαγρύπνησης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό του, οπότε κάποιες ανιχνεύσεις ενδείξεων τις έχουν ε, συμπεριλάβει στο κόστος της λειτουργίας με βάση την τωρινή ε, νομοθεσία. Οπότε δεν είναι 19, κάτι εκατομμύρια ευρώ, είναι 10, κάτι. Δηλαδή σχεδόν μείωση 50% έχουμε ε, των χρημάτων που θα πάρει ο ΕΟΦ. Ο... Το Συμβούλιο πρέπει να είναι λογικό, να μην ε, θέλει και άλλες περικοπές. Λοιπόν, αντίθετα, δεν θέλω να αυξήσω, αλλά να μειώσω το ποσό που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Και να το πω και στους κοιόδες και σε άλλους συναδέλφους. Ε, οργανώ, οργανώνω αύριο το απόγευμα μια συνάντηση με τους εμπλεκομένους στις 3.30 αν θέλετε να έρθετε συνάδελφοι να ακούσετε και τους ενδιαφερόμενους ε, να μας πούν και για τα γενώσιμα και το κατά θα πληρώνουν περισσότερο αν είναι βάση συσκευασία. Ενώ αν είναι βάση δραστικής θα πληρώνουν λιγότερο. Είναι λογικό. Θα έχουν δύο φορές μείωση. Ας το σκεφτεί η Κομισιόν να ισχύσει ε, αυτή η μονάδα και για τα γενώσιμα. Τώρα, Ντάγμαρ, που θέλει ας πούμε να δώσει κίνητρα ούτω ώστε να μειώσουν τα κράτη-μέλη το φωτοεργασία τους και να μειώσουν και το κόστος έρευνας και να αναλάβει ο ΕΟΦ. Κάποια κράτη-μέλη παραπέμπουν στο ΜΜΑ στο, τα ε, ορισμένα προϊόντα. Αλλά θα πρέπει να δούμε ε, τα προηγούμενα σκάνδαλα, όπως το Mediator. Δεν θέλουμε δηλαδή να ε, παραπέμπουν κεντρικά στο ΝΕΟΦ, γιατί αν ε, πιν, τιμωρηθούν ε, από τις, λόγω των παραπομπών που κάνουν. Σκεφτείτε τι είχε γίνει με το Mediator. Δεν υπήρχαν ε, τυπικές θεσμοθετημένες διαδικασίες ε, και ενώ συζητήθηκε πολύ δεν αντιμετωπίστηκε. Και όλοι έλεγαν δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Αυτό έγινε. Η εταιρεία το αν πέσει από κάποιες αγορές, οι Γάλλοι το άφησαν ε, τελικά έγινε γαλλικό πρόβλημα. Ε, ούτε αυτό το θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα ε, σύστημα όπου αν υπάρχει πρόβλημα να έχουμε κοινή πληροφόρηση, να την μοιραζόμαστε και να την δρούμε Εγώ μίλησα με τον ΕΟΦΕ και αυτούς που ασχολούνται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και μου λένε ότι τώρα τα κράτη-μέλη παραπέμπουν προϊόντα χωρίς τέλη. Αν είναι συνεισηγητές και ξέρω ότι άκουσα αυτό που είπε η κυρία Ροτμπέρεντ γι' αυτό, ε, για τους συζητητές. Ε, κάποιοι όμως μπορεί να έχουν όλα τα δεδομένα. Οπότε εμείς ε, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε επανάληψη εργασιών να τα ξαναμαζέψουμε. Βέβαια δεν θέλω να ε, τιμωρηθεί η παραπομπή στον κεντρικό φορέα. να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα φροντίζει να μοιράζονται τα καθήκοντα, να είναι λογικό, να αντικατοπτρίζει σωστά την κατάσταση. Υπάρχουν πολλοί σύμβουλοι εδώ που κάνουν δουλειά. Αναλαμβάνουν Μπορεί κάποιο να πει, ναι, ε, αυτό είναι ολόκληρη δουλειά, χρειάζομαι και κόσμο. Οπότε μπορεί να ε, ε, πάνε πολύ να αναλάβουν. Ε, εμείς βλέπουμε ότι ε, αναθέτει και σε εξωτερικούς ή ο ΕΟΦ, όπως στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πόσοι θα ασχοληθούν. Δεν νομίζω να είναι τόσο περίπλοκο να μην έχουμε κατά αποκοπήν ε, τέλος, το οποίο θα στηρίζεται στην ποσότητα της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Όποιος δούλεψε θα αμείβεται, γιατί τώρα η Κομισιόν επιχειρεί να πάρει τα χρήματα και να τα μοιράσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στον ΕΟΦ και να πάρουν από 50% ο καθένας. Λάθος μου φαίνεται αυτό. Όποιοι δουλεύουν θα πρέπει να αμείβονται και το ελεγκτικό συνέδριο άλλωστε αυτό περιμένει από εμά. Λογικό είναι. Ε, με το Συμβούλιο και την ομάδα εργασίας ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιες ε, έλογες αποφάσεις. Κυρία Γιάννα Κουδάκη, ο όταν ε, αρχίζα να καταπιάνομαι μου είπαν ότι είναι απλό, εόφ, ε, ε, ε, συμφωνεί, όλοι συμφωνούν. Μετά δεν συμφωνούσαν από ό,τι ε, φάνηκε, κανείς δεν συμφωνούσε με κανέναν, ούτε τα κράτη-μέλη με τον ΕΟΦ, ούτε ο ΕΟΦ με την Κομισιόν, οπότε... Περιμέναμε μετά δύο χρόνια για την πρόταση, μετά ήρθε μια πρόταση που δεν βρίσκει σύμφωνο κανένα τώρα. Πρέπει να ξαναγραφτεί, να βγει κάτι που θα βρει κάποιο Πιο σύμφωνους τέλος πάντων. Ελπίζω να ε, λειτουργήσουν όλοι με τρόπο λογικό και να προλάβουμε γιατί, όπως είπε η κυρία Ροτμπέρντ, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία, πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, να φροντίσουμε για τη χρηματοδότηση, δεν έχει νόημα να νομοθετούμε και μετά να μην έχουμε τη, τα μέσα χρηματοδότησης για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Λοιπόν, εντάξει, ε, στις 6 το απόγευμα θα είναι η προθεσμία κατάθεσης για τις 8 ενδεκάτου ε, μετά από το αίτημά σας. Στις 27-28 Νοεμβρίου θα μιλήσουμε για τις τροπολογίες και η ψηφοφορία θα γίνει 17 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας. Ενδεικτικά στην Ολομέλεια μάλλον του Απριλίου. Ε, είναι πάρα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρήσουμε. Καλώς και φτάσαμε έτσι στο τέλος της συζήτησης αυτής, αλλά δεν ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη γιατί έχουμε και την υγεία των ζώων να συζητήσουμε. Ε, η Άλτα Σούσα θα αντικαταστήσει σήμερα την Καρτίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητάει συγγνώμη η, η συγκήτρια που δεν μπορεί να είναι εδώ. Είναι βέβαια εδώ οι συνεργάτες της, θα σημειώσουν ό,τι υποθεί και θα τις μεταφέρουν ό,τι ερωτήσεις έχετε. Γι' αυτό και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα μείνω στα γενικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έκθεση αυτή. Αν δείτε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον κανονισμό αυτό για την υγεία των ζώων, το πρώτο που κοιτάει κανείς είναι ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά άρθρα. Η εισηγήτρια γνωρίζει ότι ο κανονισμός αυτός πρέπει να αποσκοπεί στο συντονισμό και την απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία των ζώων, ώστε να καταστεί λιγότερο περίπλοκη η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων. Από άποψη ουσία, ο συγκεκριμένο κανονισμό ε, περιλαμβάνει 40 διαφορετικέ ρυθμίσει όσον αφορά την υγεία των ζώων και τι περιλαμβάνει στον κανονισμό αυτό. Αλλά η συγκέντρια δεν μπορεί να καταλάβει πώ η πρόταση αυτή 262 άρθρων που πολλά από αυτά ήδη ρυθμίζονται με εκτελεστικές πράξεις, θα καταλήξουν σε απλοποίηση. Είναι μια περίπλοκη πρόταση πράγματι και η συγκήτρια έχει προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει κάποια σημεία, να τα καταστήσει πιο εύκολα κατανοητά, εξού και ο μεγάλος αριθμός τροπολογιών. Κατά τη διάρκεια ε, σύνταξης της ε, έκθεσης αυτής, η συγκήτρια έλαβε υπόψη τις δύο αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Κάτι το οποίο υπογραμμίζει την πρόληψη σε οποιαδήποτε πολιτική. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή μία υγεία, η οποία κατοχυρώνεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων του 2007 με 2013. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση απέναντι στην υγεία και λαμβάνει υπόψη τη σαφή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην υγεία και τη... των ζώων, των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στην ε, πρόταση της Επιτροπής υπάρχει η σύνδεση ανάμεσα στην υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων. Έχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ε, ζώων, όπως ανάμεσα στις ε, ασθένειες των ζώων και τις γεωργικές προ τις αγροτικές μάλλον πρακτικές μπορεί να είναι η κλωνοποίηση, η τροποποίηση του γονιώματος των ζώων, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαραγωγή τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρα και πρέπει να αναφέρονται στα άρθρα του κανονισμού αυτού. Γι' αυτό και έχει συντάξει διάφορες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση η συγκίτρια. Πάντω, θέλει επίση η συντάκτα τη νομοδότηση να τονίσει ότι γνωρίζει πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει πάνω σε ένα κείμενο για την καλή διαβίωση των ζώων, προσβλέπει σε αυτό και γι' αυτό και δεν θέλησε να προκαταλάβει τα αποτελέσματα από την πρόταση αυτή. Επιπλέον, η συντάκτα χρηματοδότηση υπογραμμίζει ότι το σημερινό σύστημα εντατική κτηνοτροφία και σημερινέ πρακτικέ περιορίζουν την κινητικότητα των ε, ζώων, κάτι το οποίο τους δημιουργεί στρες και επειδή ε, βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους τα ζώα αυτά, γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο να χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά. Κάτι το οποίο οδηγεί σε ιδεώδεις συνθήκες ε, μετάδοσης νόσων. Οπότε έτσι πλήττεται η υγεία και των ζώων, αλλά και η δημόσια υγεία. Γιατί πολύ συχνά οι ασθένειες οι οποίες απειλούν την υγεία των ζώων περνάνε όλο και περισσότερο μάλιστα στον άνθρωπο. Αν η πρόληψη αποτύχει, τότε υπάρχει κίνδυνος ξεσπάσματος ασθένειας και χρειάζονται ειδικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ολόκληρο κατάλογο με ελεγκτικά μέτρα και έχει και συντονιστικό ρόλο η συντάκτρια συμφωνεί ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμός, μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα αυτό, αλλά δεν πιστεύει ότι θα ήταν καλό να αφαιρέσουμε από τα κράτη-μέλη τη δικιά τους την ευθύνη και την δημοκρατική λογοδοσία. Η συντάκτρια πιστεύει ότι στο άρθρο 5 για τον κατάλογο των ειδικών ειδών, άρθρο 7 και η πρόληψη και ο έλεγχος που εφαρμόζονται σε ειδικέ ασθένειες, άρθρο 8, αποτελούν την ε, καρδιά, την ουσία της ρύθμισης αυτής και πιστεύει ότι αυτοί οι τομείς του κανονισμού πρέπει να υποβάλλονται σε δημοκρατικό έλεγχο, να περάσουν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και γι' αυτό για τα σημεία αυτά ε, θέλει κατεξουσιοδότηση, δεν θέλει μάλλον κατεξουσιοδότηση πράξης. Η συντάκτρια έχει συμπεριλάβει επίσης και κάποιους ορισμούς στην έκθεση αυτή για την αναπαραγωγή ιδιαίτερα. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται η κλωνοποίηση, αλλά η κλωνοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα πιο εύκολη μετάδοση ασθενειών που μπορεί να περάσουν και στον άνθρωπο και οδηγούν σε δυσμορφίες, σε διάφορα όργανα. Γι' αυτό και θέλει να υπάρξει συγκεκριμένος ορισμός. Μέχρι τώρα περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια τέτοια πρόταση για όλες τις πλευρές της κλωνοποίησης, αλλά κάθε φορά ακούμε ότι ναι, ναι, όπου να είναι θα τον έχετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως έχει εκφράσει συγκεκριμένη άποψη όσον αφορά την κλωνοποίηση και έχει πει επανειλημμένως ότι η κλωνοποίηση των ζώων με σκοπό ε, την παραγωγή τροφίμων πρέπει να απαγορεύεται. Ευχαριστώ. Πιλάρα για και μετά η Λίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση που ακούσαμε της έκθεσης της κυρίας Λεωτάρ. Όπως είπαμε και για την υγεία των φυτών, έτσι και εδώ είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώσουμε τις διάφορες ρυθμίσεις σε ένα κείμενο. Όσον αφορά τώρα τη γνωμοδότηση της κυρίας Λεωτάρ, πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται για την υγεία των ζώων προκειμένου να προλαμβάνονται οι ζωνώσεις. Δεν μιλάμε εδώ για κλωνοποίηση. Άλλες εκθέσεις αναφέρονται στην κλωνοποίηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι όλες οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τα θέματα αυτά δεν έχουν καθόλου θέση εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε νομοθέτημα για να συμπεριλάβουμε τις δικές μας ιδέες και επιθυμίες. Νομίζω ότι δεν έχει θέση εδώ λοιπόν το θέμα αυτό. Η πρόταση όντω συμπεριλαμβάνει διάφορες προβλέψεις, την επικουρικότητα για παράδειγμα με εκτελεστικέ και κατευθυντώτες πράξει. και όπως και με το προηγούμενο θέμα και εδώ είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κατάλογο των καταπροτεραιότητα στενιών στο βασικό κείμενο. Τα μέτρα επίση που πρέπει να λαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση και να συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση του κατά πόσο πρέπει να μπαίνει στον κατάλογο αυτό μια ασθένεια ή όχι. Η ελαστικότητα τώρα είναι κάτι άλλο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν ευελιξία κάθε φορά που πρόκειται για την αξιολόγηση των κινδύνων. για παράδειγμα για τους εμβολιασμού, για τις μετακινήσεις εσωτερικά μέσα σε μια χώρα των ζώων κλπ. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην επικουρικότητα. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν βέβαια οικονομικές συνέπειες. Το λένε όλοι οι φορείς και οι κτηνίατροι και δύσκολα εφαρμόζονται μερικές φορές επί τόπου είναι ένα καινούριο σύστημα που έχει μεγάλες επιπτώσεις οικονομικές αλλά και λειτουργικές για τις ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Είναι πάντως πολύ βασικό να έχουμε τη διάγνωση των ασθενειών και ο κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον μία γενική μνήμα για την ευθύνη και ποιος την έχει σε κάθε περίπτωση. Τώρα για τις ζώνες που τις έχουμε ονομάσει υποκαθεστώς ελεύθερου νόσου, προσοχή να μην έχουμε εδώ ανάλογα μέτρα και να μην δημιουργήσουμε υπερβολικό βάρος στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Τέλος, ο κανονισμός αυτός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνέπειες και γι' αυτό και πρέπει να συνδυαστεί με τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση. Το ίδιο που είπαμε και για το προηγούμενο θέμα δηλαδή. Στο άρθρο 231 αναφέρεται το σύστημα βάσει του οποίου πρέπει να εκπονήσει καταλόγους τρίτων χωρών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο σημείο 2 λέει ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν σε εθνικό επίπεδο τους καταλόγους αυτούς. Αυτό μπορεί να έχει επιπλοκές, γιατί μια χώρα μέλος μπορεί να εκπονήσει ένα τέτοιο κατάλογο, να επιτρέψει την είσοδο ενός ζώου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζώο αυτό να μετακινηθεί όμως σε άλλη χώρα, στην οποία να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει εδώ να διευκρινιστεί περισσότερο ο κανόνας. Τέλος, η ρύθμιση των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα αφιλεγόμενο ζήτημα. Είναι διμερές θέμα χωρών μεταξύ αυτού που εξάγει και αυτού που εισάγει και δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να το συμπεριλάβει σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την υγεία των ζώων. Υπενθυμίζω, πρόκειται για ένα κανονισμό υγείας των ζώων, όχι ε, καλής διαβίωσης των ζώων, οπότε η κλωνοποίηση δεν έχει καμιά δουλειά εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγιούζο η κυρία Μακάβαν και μετά ο κύριος Ζανώνη. Έχω και σχόλια από τους κοιόδης που δεν ήρθαν. Ε, την πρόταση για την υγεία των ζώων διότι εξυγχρονίζει ε, ε, οδηγίες και κανονισμούς σε ένα πλαίσιο. Το περιμέναμε καιρό για να πλουστεύσουμε το υπάρχον σύστημα. Όμως, Ανησυχούμε διότι η πρόταση θέλει να ακυρώσει ε, νομοθεσία που μόλις πριν από λίγους μήνες ε, πέρασε με συναπόφαση ε, για τη μη εμπορική μετακίνηση ζών και αναρωτιέται πώς, τι συντονισμός υπάρχει στη δουλειά της Κομισιόν. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται στο μέλλον. Η πρόταση της Κομισιόν σαφώς δεν αφορά την, υγεία, την καλή διαβίωση, αλλά την υγεία των ζώων. Αλλά η υγεία και η καλή διαβίωση είναι αλληλένδετα θέματα. Πιστεύω λοιπόν ότι για να ανταποκριθούμε στο, στην επιταγή καλύτερα πρόληψη, πρέπει να δούμε την καλή διαβίωση και να δούμε στις εκμεταλλεύσεις πώς προλαμβάνουν την κακή υγεία. Επίσης υπάρχει το θέμα της ε, μικροβιακής αντοχής ε, λόγω των αντιβιωτικών γιατί πολλά βακτήρια προέρχονται από τα ζώα. Ε, χρειάζεται λοιπόν να συνδέσουμε την υγεία των ζώων με την ανθρώπινη υγεία εδώ. μεγάλη έμφαση δίνεται στον εμβολιασμό ως εναλλακτική στη μαζική θανάτωση ζώων σε περίπτωση ε, ζωνώσεων. Η, κοινότητα, η, κοινωνία γίνεται λιγότερο ανεκτική στην θανάτωση. Και η συγγήτρια αναφέρεται σε περιβαλλοντικά θέματα πέρα από την ε, μαζική θανάτωση ζώων. Το άλλο που θέτει ο σκιώδης συγητής είναι το θέμα των εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων. Κάποιες είναι σημαντικές και ουσιαστικές, αλλά θέλει σαφή οδικό χάρτη ε, ε, σχετικά με το τι εξουσιοδοτούμε και χρονοδιαγράμματα που σχεδιάζονται και οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν με το Κοινοβούλιο. Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα σε όλα αυτά. Βέβαια, το πρόβλημα της υγιεινής του κρέατος προέκυψε το καλοκαίρι με τις, εκτελεστη... με τις κατεξουσιοδότηση πράξη, ε, που έπρεπε να εξετάσουμε και να ελέγξουμε μόλις γυρίσαμε πίσω από τις διακοπές. Στο μέλλον λοιπόν όταν εξετάζει η ε, κατεξουσιοδότηση πράξης η Κομισιόν πρέπει να δίνει και χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή το 2014 θα υπολογίζουμε να έρθουν αυτές. Όπως έχουμε και εμείς χρονοδιάγραμμα. Όχι να μας τις πετάνε στο κεφάλι και να μας λένε έλα κοινοβούλιο στα σβέλτα ε, να δουλέψετε. Θέλουμε χρονοδιάγραμμα λοιπόν όπως έχουν και εκείνοι και ε, όποτε παραβιάζεται το χρονοδιάγραμμα να το εξηγούν κιόλα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέας Ζανώνη και μετά η κυρία Άννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση κανονισμού αφορά την υγεία των ζώων, άρα είναι μια πρόταση πολύ σημαντική γιατί καταργεί 40 περίπου κανονισμούς και οδηγίες που αφορούν την υγεία των ζώων ακριβώς. Παρόλο που θεωρούμε τον κανονισμό αυτό, τον καινούριο κανονισμό, πολύ πολύπλοκο και καλά ε, διαρθρωμένο όσον αφορά την υγεία των ζώων, ε, σίγουρα θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει στενή σχέση, άμεση σχέση, ανάμεσα στην υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων. Άρα η υγεία των ζώων συσχετίζεται άμεσα με την καλή διαβίωση των ίδιων των ζώων και μεταξύ άλλων είναι η εγγύηση και για τον καταναλωτή. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ε, δεν υπάρχει υγεία των ζώων πολύ συχνά λόγω μη καλής διαβίωσης των ζώων, ε, τότε δημιουργούνται προβλήματα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές ασθένειες που μπορεί να έχουν συνέπειες και για την ανθρώπινη υγεία. Πολύ συχνά αναφέρεται το παράδειγμα ε, της, ε, της ασθένειας των τρελών αγελάδων ή την γρήπη των πτηνών που στην βορειοανατολική Ιταλία είχαμε ε, και ανθρώπινα ε, θύματα λόγω της ε, γρήπης των πτηνών. Άρα ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ιδιαίτερα ε, μεγάλες και έντονες προσπάθειες όπου αυξάνονται οι παράγοντες κινδύνου. Τώρα υπάρχουν κάποιες επιμέρους διατάξεις, παραδείγματο χάρη όσον αφορά τις επεμβάσεις επί των αγρίων ζώων. Κατά τη γνώμη μου δεν λαμβάνεται ε, δεόντως υπόψη το θέμα της ε, διατήρησης των άγριων ζώων ε, γίνεται γενικά λόγος για καταπολέμηση των ασθενειών, των επιδημιών κλπ. Δεν αναφέρεται όμως πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε ε, απέναντι στα άγρια είδη που μπορεί να έχουν προσβληθεί ή που μπορεί να συμβάλλουν στην εξάπλωση συγκεκριμένων ασθενειών. Και για το σημείο αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Μετά, και πάλι για τα άγρια ζώα, ε, θεωρώ ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει μια νομική πλαισίωση για την προστασία των ε, αγρίων ε, ειδών, μια ειδική τέτοια νομοθεσία. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία θεωρούνται κληρονομιά του κράτους, η άγρια πανίδα δηλαδή. Γι' αυτό αυτές οι λεπτομέρειες θα πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα μέσα στην πρόταση. Οι καταναλωτές τώρα ε, θεωρώ ότι παρακολουθούν με προσοχή την πρόταση αυτή γιατί αυτή η πρόταση για την ε, υγεία των ζώων κατά τη γνώμη μου ε, προϋποθέτει και κάποια πρότυπα, κάποια στάνταρα όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, διότι όταν έχουμε υγιή και με καλή διαβίωση ζώα, έχουμε και πιο ασφαλή και καλύτερα προϊόντα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, παραδείγματο χάρη για κάποιες ανησυχίες που εκφράζει σχετικά με την κατάργηση ε, της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοηδών και την σήμανση του βοήου κρέατος. Είναι σίγουρα σημαντικό να γνωρίζουμε ε, όλα τα, όλη την πορεία που ακολουθεί ε, ε, ένα προϊόν και όσο μεγαλύτερη χνηλασιμότητα υπάρχει τόσο το καλύτερο. Άρα το σημείο αυτό θα πρέπει να εφαρθεί κατά τη γνώμη μου. Ε, χρειάζεται να υπάρχουν έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια της ε, αλυσίδας από την εκτροφή μέχρι τη μεταφορά και στη συνέχεια. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός άρθρων που προβλέπουν μεγάλες εξουσίες της Κομισιόν με πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Ε, όμως για ορισμένα σημεία ε, ο κίνδυνο είναι ε, σε σχέση με την νομοθεσία αυτή να μην ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι το περιεχόμενο που μπορεί να μας ενδιαφέρει και να μας αφορά. Και μετά υπάρχουν και πολλές παρεκκλήσεις, πολλές εξαιρέσεις όντως. Υπάρχουν πολλά συστήματα αυτοπιστοποίησης. Ίσως θα ήταν να αξιοποιηθεί καλύτερα ο ρόλος των ε, κτηνιάτρων όμως, αντί να τους αφήνουμε έτσι ε, στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο. Ε, υπάρχουν επίσης κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων, γιατί προβλέπονται εκεί διάφορες εξαιρέσεις και υπάρχουν και κάποιες απαλλαγές όσον αφορά την υποχρέωση ε, εγγραφής σε Μητρώα σε σχέση με τις διάφορες εγκαταστάσεις. Γενικά μπορώ να συμφωνήσω με την ε, γραμμή που υιοθέτησε η συγγήτρια και από το μεγάλο αριθμό των τροπολογιών, ας μην το ξεχνάμε αυτό, ε, που είναι 189, πολλές από αυτές θεωρώ ότι βελτιώνουν την πρόταση. Να μην ξεχνάμε ότι η πολυπλοκότητα αυτής της νομοθεσίας ε, απαιτεί ευάθυνση πολύ μεγαλύτερη. Γιατί πραγματικά όταν προσπαθούμε να, να συνθέσουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα ενιαίο κείμενο... Ε, διατάξεις που προέρχονται από 40 διαφορετικά νομοθετήματα, ε, πραγματικά υπάρχει κίνδυνος κάτι να χάσουμε σε αυτή τη ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Ιάννα Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ την ε, εισηγήτρια που δεν είναι σήμερα εδώ και που άρχισε έγκαιρα τη δουλειά της ως εισηγήτρια. Για μένα το θέμα είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πραγματικά που επιτέλους αρχίσαμε να το επεξεργαζόμεθα. Ξέρω ότι αυτή είναι, αυτός είναι ένας κανονισμός για την υγεία των ζώων, αλλά τα ζώα είναι καλά και υγιή όταν διαβιώνουν καλά και δεν έχει και η συνάδελφος από το ΕΛΚ. Κυρία Γιούζο, τα υγιή ζώα σημαίνει ε, ότι θα τρώμε και εμείς καλά. Και η καλή προστασία των ζώων συμβάλλει σε αυτό. Προστασία των ζώων πολύ σημαντική λοιπόν. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε μια ένεση και να τελειώνει το θέμα ή να περιοριζόμαστε σε έναν εμβολιασμό δεν έχουμε την ίδια άποψη. Έτσι όπως βλέπω τα κείμενα. Αλλά για, μας, για μένα είναι σημαντικό τα ζώα να αντιμετωπίζονται με βάση κανόνες για την προστασία τους. Είτε πρόκειται για τη μεταφορά, είτε για ε, οτιδήποτε άλλο. Είναι όλα αυτά σημαντικά για την ποιότητα του κρέατος που θα φτάσει στο πιάτο μας. Είμαι ευγνώμων στην εισηγήτρια σχετικά με την αντίληψη μία υγεία, One Health Concept και για μένα είναι σαφώς ότι τα καλά τρόφιμα προέρχονται από υγιή ζωά. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα για μένα της υπερβολικής αντιβίωσης και της προληπτικής αντιβίωσης που χορηγείται πολλές φορές στα ζώα. Και βέβαια είναι καλό ότι κάποιες νόσοι, ζωονόσοι, όπως η νόσος των τρελών αγελάδων, η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια των βοηδών αναφέρεται εδώ. Και βέβαια το θέμα είναι πόση ισχύ θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα αναθέτει σε άλλους. Πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη, γιατί έτσι θα βρούμε που ε, ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές. Είναι καλή η περίπτωση αυτή. Λοιπόν, τελειώσαμε με τους σκιώδεις. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οι δύο ομιλητέ που απομένουν, η συνάδελφο Λούψεβα και η ε, κυρία Σνέλχαρτ και η κυρία Αγιούζο, που θέλει να απαντήσει, θα πάρουν από ένα λεπτό η ε, κάθε μία. Η κυρία Σνέλχαρτ θα τα καταφέρει. Η κυρία Λούψεβα όμω προηγείται. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω βουλγαρικά κύριε Πρόεδρε εγώ υποστηρίζω δύο σημαντικές ιδέες σε αυτή τη γνωμοδότηση. Πρώτον, καλύτερα η πρόληψη από τη θεραπεία, πολύ σημαντική η έμφαση εκεί και τέλος το συμπέρασμα στο σχέδιο γνωμοδότησης για την ε, πρακτική της μαζικής θανάτωσης ε, που θα πρέπει να ε, χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στα κάτωθη. Πρώτον, διασυνοριακή μεταφορά, μετάδοση νόσων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν η ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν λειτουργεί, αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Στη δική μου την περιφέρεια πριν από τρεις εβδομάδες πάνω από 200 ζώα θανατώθηκαν λόγω μετάδοσης νόσου από την Τουρκία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο ακριβή και συγκεκριμένη ρύθμιση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση. Ε, χρειαζόμαστε μέτρα συγχρονισμού για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Και ε, να καταφέρουμε να αποφύγουμε την μαζική θανάτωση. Τέλος, ε, η έγκριση των εμβολίων και των εμβολιασμών. Θα πρέπει να επιτρέπονται εμβολιασμοί σε περίπτωση όπου είναι αναγκαίοι στις ε, παραμεθόριες περιοχές. Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να συμβαδίζουν, να συνοδεύονται από ε, στοιχεία σχετικά με περιοχές ελεύθερες νόσου. Ο κύριος Νέλχαρτ, ε, θα είμαι σύντομος, δεν έχουμε χρόνο. Η πρόταση αυτή συζητείται εδώ και καιρό. Το 2007 μέχρι το 2013 μιλάμε για τη στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά αναφέραμε γενικά που εστιάζονται τώρα εδώ συγκεκριμένα. Έχω ένα πρόβλημα όμως γιατί στην πρόταση αυτή ε, περιλαμβάνονται παράγραφοι που πρέπει να ε, αναφέρονται στη δέσμη μέτρων για την υγεία, για τα οικόσιτα ζώα κλπ. Αυτά έχουν ρυθμιστεί και βλέπω εδώ ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει ακόλουθες δραστηριότητες και μετά αναφέρεται και η κατεξουσιοδότηση πράξης κομισιών. Τώρα, εμείς ε, είχαμε εγκρίνει εδώ και χρόνια κανονισμούς που λειτουργούν. Αυτούς δεν τους λαμβάνει υπόψη κομισιόν. Ε, υπάρχει ένα σύστημα λειτουργικό. Βεβαίω είναι ευρύτατο, έχουμε 50 βασικές ε, οδηγίες που εδώ θα συγχωνευτούν. Αλλά εις ό,τι αφορά τώρα τα 20 τα ζώα βλέπουμε άλλη προσέγγιση. Δεν λέει τι πρέπει να γίνεται, πράγματα που τα είχαμε αποφασίσει, γιατί σε τρεις συνεδριάσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σακωνόμαστε σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να είναι η κατεξουσιοδότηση πράξη. Τα συμφωνήσαμε και τώρα δεν ισχύει πια αυτό. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Ε, είναι πραγματικά πρόκληση αυτό που γίνεται, το λέω στην Κομισιόν μέσα από τις κατεξουσιοδότηση πράξης για τη χρηματοδότηση. Οι περισσότεροι είπαμε, είπαν ότι δεν θέλουμε εκτελεστική πράξη για τις ζωνόσους. Ε, είπαμε ότι θα πάρουμε τις κατεξουσιοδότηση. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να δείξουμε ποια είναι τα όρια στην Κομισιόν τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Έτσι δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει ανασφάλεια δικαίου μεταξύ των χρηστών. Οπότε δεν μπορεί να περάσει αυτό το σύστημα. Ε, θα πρέπει να ασκήσουμε περισσότερες πιέσεις. Ε, μίλησε λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ε, η Κρίστα θα μιλήσει λιγότερο τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Γιούζο. Θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είμαι κατά της, διαβίωσης, της καλής διαβίωσης των ζώων κάθε άλλο. Απλώς έχουμε ρυθμίσεις για την καλή διαβίωση των ζώων. Το να βάλουμε εδώ. Αυτά τα οποία θα βάλουμε στον άλλο κανονισμό, θα είναι υποχρεωτικά, είναι περιττό. Εξάλλου βαραίνουν πάρα πολύ το κείμενο με θέματα τα οποία δεν είναι ο πραγματικός μας στόχος. Εδώ ο στόχος μας είναι η υγεία των ζώων. Τελεία. Ευχαριστώ και τώρα η Κομισιόν που απαντήσει στις επικρίσεις. Εδώ λέμε ότι είναι πρόκληση αυτό η πρότασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί τελείωσε ο χρόνος. Θα ήθελα να ανακεφαλαίωσω λιγάκι. Αυτό που προτείνουμε εδώ είναι μια εντελώς νέα νομοθεσία η οποία καλύπτει 40 χρόνια νομοθεσίας για την υγεία των ζώων από τα τέλη της δεκαετίας του 60 που ξεκίνησαν οι πρώτοι κανονισμοί του Συμβουλίου, μετά Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, που κάλυπταν όλα τα θέματα της υγείας των ζώων. Και ενώ ε, βέβαια μεταδοτικές ε, ασθένειες των ζώων. Μόνο για μεταδοτικές ζωονόσους μιλάμε. Όλες αυτές οι νομοθεσίες λοιπόν και οι πιο πρόσφατες θα καλυφθούν από αυτόν τον νέο κανονισμό. Θα επανέλθω σε αυτά που ανέφερε μόλις ο δόκτωρ Σενέλε. Δηλαδή ότι ακόμα και οι πιο πρόσφατες νομοθεσίες που οδήγησαν σε μακροχρόνιους τριλόγους κλπ θα θυμάστε τον τελευταίο, και αυτά τα τελευταία νομοθετήματα θα καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι σαφές και να ε, ξεκαθαριστεί. Ε, το, το δηλώνει σαφώς η Κομισιόν. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε στον τριμερή διάλογο και το ανέφερε ο Επίτροπος προς τους Ευρωβουλευτές. Γράφει, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ε, πρόσφατες ε, νομοθετικές συμφωνίες για τα ζώα συντροφιάς και για τη σήμαση των βοηδών θα ε, υπάρχουν μέσα στη νέα πρόταση της Κομισιόν. Δεν θα υπάρχει λοιπόν καμία αλλαγή σε σχέση με αυτά που συμφωνήσαμε εδώ μετά από μακροχρόνιο τριμερή διάλογο. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα νομοθεσία που συνοψίζει 40 οδηγίες και εκατοντάδες εκατοντάδων εφαρμοστικών αποφασίσεων της Κομισιόν. Ναι, είναι τεράστιο λοιπόν το νομοθέτημα, αλλά επίσης μειώνει τον αριθμό των εξουσιών που ανατίθεται στην Κομισιόν. Τώρα, αν αφαιρέσουμε κάθε εξουσία από την Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 800 τέτοιε εξουδοτήσεις. Μετά την νέα νομοθεσία θα είναι μόνο 160. Βλέπετε λοιπόν πόσο μειώνεται ε, ο αριθμός των ε, εξουδοτήσεων. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η πρόταση αυτή δεν αφορά την κλωνοποίηση, η πρόταση δεν αφορά την καλή διαβίωση των ζώων και επίσης δεν αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς την κλωνοποίηση, μπορώ να επαναλάβω αυτά που είπαμε νωρίτερα, θα υπάρξει μια ε, συνάντηση με ε, θα υπάρχει μια ε, ειδικά προγραμματισμένη ε, σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το Νοέμβριο για την κλωνοποίηση και μόλις ληφθεί η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Για την καλή διαβίωση των ζώων επίσης δεν καλύπτεται αυτή την πρόταση όπως είπα. Είναι μια άλλη διαδικασία πάλι που επίσης ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και η οποία θα οδηγήσει με συνεχιζόμενη εργασία που πραγματοποιείται στις υπηρεσίες της Κομισιόν και θα συνεχίσει να εξελίσσεται όπως προβλέπεται η εργασία αυτή. Τώρα, για τον, το θέμα του καταλόγου των ασθενειών και του καταλόγου των ειδών που ανέφεραν αρκετοί ευρωβουλευτές, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ουσιαστικό τμήμα αυτής της πρότασης. Τα κριτήρια για την καταλογοποίηση των ασθενειών ε, υπάρχουν μέσα στην ε, πρόταση. Πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει αντίκτυπος για, την, ε, για τον ζώο, ότι υπάρχει πρόβλημα με το εμπόριο κλπ. Πρέπει να είμαστε όμως ευέλικτοι. Θυμάστε το πρόβλημα τη γλουτένη που προέκυψε πριν από τρία χρόνια. Αν δεν ήμασταν αρκετά ελαστικοί, δεν θα ήμασταν σε θέση να προτείνουμε κανόνες για το εμπόριο της γλουτένης και δεν θα μπορούσαμε να εξοδέψουμε 180 εκατομμύρια τον χρόνο για να, όχι για τη γλουτένη, για ένα άλλο πρόβλημα, δεν θα μπορούσαμε να ε, εξοδέψουμε 180 εκατομμύρια για τον εμβολιασμό των ζώων για το πρόβλημα αυτό. Ε, τώρα, για τις ε, εξαιρέσεις, όταν υπάρχουν πήγουσες συνθήκες, όταν είμαστε σε κατάσταση κρίσης, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Και αυτό το τοποθετούμε μέσα στο κείμενο. Ε, παραμένουν εξαιρέσεις αυτά. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά μην ξεχνάτε τι έγινε το 2001 με τον Αυτόδη πυρετό, οπότε χρειάστηκε να σφάξουμε εκατομμύρια ζώα, να θανατώσουμε εκατομμύρια ζώα, ε, έπρεπε να είμαστε θέση να δουλέψουμε αποτελεσματικά. Και αυτή την ευελιξία θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Επίσης, έγιναν κάποιες αναφορές στην αντοχή στα αντιβιωτικά. Ε, υπάρχουν παθογόνα που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά και καλύπτονται από αυτή την πρόταση. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν ειδικά. Αυτές ήταν ε, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω απαντώντας στις διάφορες παρατηρήσεις των ε, Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και για την κλωνοποίηση θα πάρουμε πρόταση. Ένα είναι σαφές η πρόταση της Κομισιόν αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται ε, των αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου που διεκόπη. Ε, αυτά τα συζητήσαμε με τους συντονιστές, ε, οτιδήποτε άλλο θα ήταν οπισθοχώρηση. Έτσι θα ήθελα και εγώ να το τονίσω αυτό, ότι υπάρχει συμφωνία διαπαραταξιακή. Όλες οι ομάδες συμφωνούν ότι περιμένουμε για την κλωνοποίηση πρόταση, που δεν θα υπολείπεται αυτής. Δεν ήταν όμως αυτό το θέμα σήμερα, το, θέμα ήταν η υγεία των ζώων σήμερα. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και σχεδόν τελειώσαμε. Α, 21 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 16-17 θα ψηφίσουμε εδώ στην Γεωργία το Φεβρουάριο και Μάρτιο-Απρίλιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Λοιπόν, κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα εμείς θα ξαναειδωθούμε στις 7 Νοεμβρίου πάλι, σε δύο μέρες δηλαδή. Κοινή συνεδρίαση Ήτρε και Ένβη. Από τις 9 μέχρι τις 12.30 ε, θα χαρώ να δω πολλούς συναδέλφους. Στις 14 Νοεμβρίου είναι η μίνι συνεδρίαση που αρχίζει στις 9 και πρόκειται για τη Μαγιώτε, 30 λεπτά ε, κατά μέγιστον, γιατί έχουμε μεγάλη χρονική πίεση, στις 27, και αυτό είναι εξαίρεση, γιατί δεν θα είναι μια πολιτική ομάδα παρούσα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. 27 Νοεμβρίου και 28 Νοεμβρίου, ως ήθιστε 9 με 12,5 και 3 με 6,5 θα γίνει η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Καλή σας όρεξη και θα σας δω φαντάζομαι κάποιους από εσά τους τριμερείς διαλόγους γιατί γίνονται παράλληλα πολλές. Πολλοί. Και ε, ορισμένοι θα πάνε κατευθείαν να συναντηθούν στην συνεδρία των σκιωδών.